Και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, η ίδια η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής θα είναι αρκετά σύντομη. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τη Ζανίν Χένις πρώην συνάδελφό μας, η οποία επιστρέφει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευχαρίστηση, ελπίζω. Είναι ε, υπουργό Άμυνα, πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση. Συγχαρητήρια εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε την χαρά και την τιμή να έρθετε στην Υποεπιτροπή η οποία πριν από το Συμβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου αφιερωμένη στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα προσπαθήσει να ακούσει όσο το δυνατόν περισσότερους υπουργούς των κρατών μελών. Όλοι δεν προσέρχονται. Ευχαριστώ που δεχτήκατε. Οι κάτω είναι ένας πρωταγωνιστής σημαντικός ε, στο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σκέλος της πολιτικής αυτής. Ήμουνα με τον συνάδελφο Λίμπερμαν στην Καμπούλ και είδαμε την σημασία ε, των στρατευμάτων ε, των Ολλανδικών. Οι κατοχώρες επίσης θα αναπτυχθούν στο Μαλί οι δυνάμεις των κατοχωρών, οι κατοχώρες θα συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και είναι και μια χώρα η οποία είναι σε φάση εχμής ως προς την αμοιβεοποίηση, ως την αποκοινού ε, ανάληψη ε, με, την, με το Βέλγιο, με την Γερμανία για θαλάσσιες μονάδες ε, και είσαστε αρκετά προχωρημένοι σε σχέση με το ευρωπαϊκό κίνημα Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους ε, για τους οποίους νομίζουμε ότι η συζήτηση αυτή θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και συνοπτικοί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Uh, Ήμουν για έξι χρόνια μέλος εδώ έφυγα από το Κοινοβούλιο το 2010 και το ότι είμαι μαζί σας σήμερα ε, μου θυμίζει πολύ καλά πράγματα. Πριν γίνω βουλευτής είχα περάσει αρκετά χρόνια στην ε, Λετωνία, στη Ρήγα, σαν ε, υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ήταν ακόμα μέλος. Η Λετωνία ήταν μια χώρα που προσπαθούσε να κάνει την περίοδο της μετάβασης και ζώντας εκεί μου απέδειξε ότι η ευημερία και η ελευθερία δεν είναι τίποτα το δεδομένο. Κατέληξα λοιπόν ότι ένα ασφαλές περιβάλλον σαν και αυτό στο οποίο μεγάλωσα δεν είναι κάτι το προφανές και αξίζει να πολεμάει κανείς γι' αυτό σε καθημερινή βάση. Αρκετά χρόνια αυτή, μετά αυτή η ιδέα μου, έκανε, μου ξανάρθε αν θέλετε μετά από τις επισκέψεις που έκανα στη Λευκορωσία. Μόλις έφτασα εκεί δεν είδα την αντιπολίτευση και μου απαγόρευσαν την, την είσοδο οι εκπρόσωποι του Λουκασένκο και του καθεστώτος του και αυτό είναι κάτι το οποίο μου ενίσχυσε την αντίληψη ότι η Ευρώπη έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και πρέπει να υποστηρίξουμε τη μάχη για τη δημοκρατία στη Λευκορωσία. Η σταθερότητα και η δημοκρατία σε χώρες όπως η Λευκορωσία δεν ωφελούν μόνο τους πολίτες αυτών των χωρών, αλλά είναι και προς όφελος της ιδείας της Ευρώπης. Όλοι τώρα πλέον συζητάμε ότι γεγονότα σε άλλα μέρη του κόσμου, κοντά ή πιο πιο μακριά επηρεάζουν άμεσα την ευημερία μας και την ασφάλειά μας. Η ευρωπαϊκή εμπλοκή σε περιφερειακές σειράξεις όχι μόνο προσπαθεί να ε, μειώσει τις εκδηλώσεις τρομοκρατίας, αλλά να διασφαλίσει και την προμήθεια ε, εμπορικών προϊόντων απαραίτητων για την ανάπτυξή μας και κυρίως πρώτων υλών. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς εστίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και συνεχώς μετακινούνται και κάθε φορά ο άνεμος αλλάζει ταχύτητα και κατεύθυνση. Το συνολικό γεωπολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερος ρευστό. Η ισορροπία δυνάμεων μετακινείται συνεχώς και νέοι ε, πρωταγωνιστές αποκτούν μεγάλη σημασία. Τίποτα δεν είναι πλέον τόσο προβλέψιμο. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι η αβεβαιότητα είναι το ισχυρότερο χαρακτηριστικό των διεθνών σχέσεων. Είμαι πεπισμένη πάντως πως σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες και τις αναδιόμενες απειλές μόνο με συνεργατικό τρόπο. Απαιτείται πιο δραστήρια, πιο συνεκτική και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας πρέπει να αναλάβουμε το δικό μας βάρος και πρέπει να αναλάβουμε και τους κινδύνους. Αυτό θα στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Ηνωμένε Πολιτείε τον απαραίτητο εταίρο μας στον τομέα της ευρωπαϊκής ασφάλειας για 65 ολόκληρα χρόνια. Στο παρελθόν υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μια ισχυρή Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει εναντίον του ΝΑΤΟ. Όχι βέβαια, είμαι πεπισμένη ότι θα ενισχύσουμε έτσι τις διατλαντικές μας σχέσεις και δεν θα πρέπει βέβαια να ζητάμε τις επικαλύψεις, ούτε θα προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά να διασφαλίσουμε τη συνεργασία, το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ότι τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας έχουν ρόλο και σημασία. Πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρώπη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γίνει ένας αξιόπιστος παροχέας ασφάλειας και στην περιοχή και πέραν αυτής. Σήμερα, λίγες εβδομάδες από αυτή τη σημαντική συνάντηση του Συμβουλίου, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν ακολουθούμε τον σωστό δρόμο. Έτσι νομίζω. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη για επιτάχυνση των προσπαθειών μας. Είναι πλέον καιρός η συνεργασία μας να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Αυτό ισχύει κυρίως για τη στρατιωτική μας συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα η δημοσιονομική θα παραμείνει μαζί μας για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας και να πετύχουμε τις οικονομίες κλίμακας που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη στρατιωτική μας αποτελεσματικότητα. Παράλληλα θα πρέπει με σοφό τρόπο να δαπανούμε τα χρήματα των φορολογουμένων μας. Πάντως οι ελλείψεις οι στρατιωτικές του ΝΑΤΟ που φαίνονται και στο ΝΑΤΟ και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με κοινό τρόπο μπορεί να καλυφθούν. Αυτό σημαίνει καλύτερη και στενότερη πολιτική συνεργασία. Δεν θα πρέπει οι χώρες να λειτουργούν η μία εναντίον της άλλη αλλά συμπληρωματικά. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την δυνατότητα παρέμβασής μας, αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και τότε μόνο μπορούμε να πούμε ότι οι πράγματι πιστεύουμε στην ΚΕΠΑ. Και τότε μόνο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας αξιόπιστος παροχέας ασφάλειας και τότε μόνο η Ευρώπη θα είναι ένας αξιόπιστος και ικανός σύμμαχος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα ευρωπαϊκό στρατό ή ένα στρατό του ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη, οι συνδυασμοί κρατών μελών θα πρέπει να παρέχουν στην Ευρώπη με τα στρατιωτικά μέσα τα οποία έχει ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρωπαϊκό έθνος είναι και απαραίτητο και υπεύθυνο για τα θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όπως ε, είναι γνωστό από παλαιόθεν, ε, πράγματι όλοι για έναν και ένας για όλους. Ε, έχουμε επίσης και την πρόσφατη έκθεση της Lady Ashton σχετικά με τις ομαδοποιήσεις ε, στις οποίες πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ε, για να βελτιώσουμε την ΚΕΠΑ. Φαίνεται μέσα από την έκθεση ότι έχουμε ελλείψεις και σε επίπεδο ικανοτήτων και σε επίπεδο συνεκτικότητας για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, συγκεκριμένοι, να χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν και δεν μπορώ πάμε να συμφωνήσω με αυτή τη λογική. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα στρατηγία, δεν χρειαζόμαστε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους και περισσότερη γραφειοκρατία. Απαιτείται όμως ηγετική ικανότητα, αφιέρωση στην προσπάθεια και θάρρος. Εκ των κάτω θα πρέπει προφανώς να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σας έλθω τώρα σε κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα της έκθεσης. Καταρχάς, η συνολική αντιμετώπιση, αν θέλετε. Η Ολλανδία υποστηρίζει την σωστή χρήση των υπαρχόντων μέσων, αν θέλετε. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα σε χώρες που αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Και ελπίζω ότι είπατε η εκπρόσωπος θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ε, γρήγορα σχετικά με τους ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς σχηματισμούς. Είπα, χρησιμοποιήστε τους ή θα τους χάσετε. Προφανώς οι σχηματισμοί αυτοί ήταν και εξακολουθούν να είναι σημαντικοί για να διασφαλίσουν τη διαλετουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών. Αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί όσο τουλάχιστον γίνεται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν παράδειγμα στην αρχή μιας εκπαιδευτικής αποστολής, παρέχοντας προστασία των δυνάμεων. Γιατί να μην χρησιμοποιεί λοιπόν τις σωστά εκπαιδευμένες και διαθέσιμες τέτοιες στρατιωτικές δυνάμεις. Βέβαια, η διαδικασία λήψεως αποφάσεων είναι αργή και απαιτεί πάρα πολύ ε, προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν αυτά να προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε όπως και σε επίπεδο σενάριων, σενάριων συγγνώμη, και πρέπει οι διαβουλεύσεις να εντατικοποιηθούν. Οι πέντε χώρες που συνεισφέρουν στο στον ευρωπαϊκό σχηματισμό του οποίου ηγείται το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Λετωνία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν γίνει προτάσεις έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, κοινέ ασκήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινέ λήψεις αποφάσεων, τακτικές διαδικασίες πιστοποίησης των σχηματισμών μάχης, όπως επίσης και συγκεκριμένα ε, ε, προγραμματικά σενάρια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου σε κάποιες αποφάσεις που θα συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση των ικανοτήτων θα πρέπει νομίζω να είναι ο βασικός στόχος της έκθεσης. Όπως είπα, οι ελλείψεις οι στρατιωτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διορθωθούν μέσω κοινών αντιλήψεων και δράσεων. Η έκθεση της Lady τον υποστηρίζει πάρα πολύ σωστά ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται τις ικανότητες οι οποίες υπάρχουν. Αυτό σημαίνει νέος προγραμματισμός στον τομέα ακριβώς ε, της σχεδίασης, της απόκτησης, ε, της εκπαίδευσης και της επιμελητίας αν θέλουμε πράγματι να είμαστε σοβαροί σε σχέση με την κάλυψη των κενών της στρατιωτικής ικανότητας της Ευρώπης, θα πρέπει να σταματήσουμε ε, την πρακτική που ισχύει, η οποία στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να ε, προκαλεί την εθνική εσωστρέφεια. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα των ικανοτήτων δεν είναι μια επιλογή την οποία θα πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Έχει πάρα πολύ σημασία να δράσουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα ακριβώς με τον κώδικα συμπεριφοράς συνδυασμού δυνάμεων και διαμήρασης δυνάμεων. Αυτό θα επιτρέψει να δημιουργούνται ικανότητες με αποτελεσματικό τρόπο, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων δυνάμεων. Θα πρέπει φυσικά να συνεχίσουμε να είμαστε διαλειτουργικοί όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και με τους εταίρους μας και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι 28 χώρες θα πρέπει να κάνουν πάντα το ίδιο πράγμα, όχι βέβαια. Όπως είπα, ε, μια διαδικασία εκ των κάτω προς τα πάνω με ικανή διακυβέρνηση εκ των άνω προς τα κάτω είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Αυτό περιλαμβάνεται και στην έκθεση της Λέντιάστον. Θα πρέπει με μικρές ομάδες να προχωρήσουμε που θα εμπλέκονται φυσικά και τα 28 κράτη-μέλη. Οι ικανότητες ε, σε μικρές ομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εμπνεύσουν άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Η συνεργασία αυτή μπορεί να ανοίξει σε μια ιστερότερη φάση και σε άλλα κράτη-μέλη. Η συνεργασία της χώρας μου, σαν παράδειγμα με το Βέλγιο, έχει οδηγήσει σε πλήρως ενσωματωμένα και ολοκληρωμένα ναυτικά, πολεμικά ναυτικά. Η Ολλανδία συνεργάζεται επίσης με τη Γερμανία και το γερμανικό-ολλανδικό ε, κοινό στρατιωτικό σώμα. Έχουμε ένα μόνιμο στρατηγείο. Έχουμε επίσης υπογράψει και μία επιστολή προθέσεων με τον ομόλογό μου του Βελγίου για, μια, για έναν προγραμματισμό αεροπορικών περιπολιών. Και υπάρχει επίσης και η αμφίβια στρατιωτική δύναμη Ηνωμένου Βασιλείου Ολλανδίας. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα από ένα μακρύ κατάλογο πρωτοβουλειών συνεργασίας. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια κρίσιμη πλευρά στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία είναι η κατανόηση ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εφόσον οι εταίροι είναι έμπιστοι και προβλέψιμοι στι δράσει του. Το να λέει κανεί ναι στη στρατιωτική συνεργασία σημαίνει ότι λέει ναι στη στρατιωτική συνεργασία. Οι αξιόπιστοι εταίροι σε καμία περίπτωση δεν παίρνουν πίσω τις δυνάμεις του την τελευταία στιγμή. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πολιτικό κενό και θα απειλήσει τις στρατιωτικές συνεργασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει όμως γίνει απόλυτα ακόμα δεκτό. Είναι απαραίτητο τα μέλη του σώματος όπως επίσης και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να εμπλακούν με ουσιαστικό τρόπο στη συζήτηση που προηγήθηκε και αυτό είναι το σημείο στο οποίο οι επιτροπές σας θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο διευκολύνοντας τακτικές μορφές συνεργασίας ανάμεσα στα κοινοβούλια. Είμαι πεπισμένη ότι ο διαφορετικός διάλογος θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Όταν πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας, να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να βελτιστοποιήσουμε τις κοινέ μας ενέργειες, αυτό θα γίνει όταν όλοι νιώθουμε με τον ίδιο τρόπο εμπλεκόμενοι. Και απαιτείται φυσικά και δημόσια υποστήριξη. Όμως, η στενή στρατιωτική συνεργασία γίνεται αντιληπτή από πάρα πολλούς σαν ένας περιορισμός σε επίπεδο κυριαρχίας και εθνικού ελέγχου και ε, σαν αποτέλεσμα αυτού πάρα πολλές φορές υπονομεύουμε οι ίδιοι την αποτελεσματικότητά μας και την αποδοτικότητά μας. Όμως αν θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας μέσω στρατιωτικών μέσων η συνεργασία είναι απαραίτητη. Και αν θεωρούμε ότι οι στρατιωτικές μας δυνάμεις μπορεί να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα βελτιώσουμε την ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε σε περιόδους κρίσης. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή συνεργασία στο στρατιωτικό τομέα δεν είναι ένας περιορισμός, αλλά μια βελτίωση της προστασίας της κυριαρχίας μας και της ασφάλειάς μας. Υπερασματικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Κατανοούν ότι υπάρχει ανάγκη η Ευρώπη να γίνει ένας αξιόπιστος παροχέας ασφάλειας και στην άμεση περιφέρεια αλλά και πέραν αυτής. Πρέπει να αναιρεθούν λοιπόν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια απαιτείται μια πιο συνεκτική και ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Βοηθήστε προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω το μήνυμα που σας μετέφερα να το μεταδώσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Bien, merci euh, Euh, Ευχαριστώ πολύ ε, για αυτήν την παρουσίαση, η οποία ήταν πάρα πολύ ρεαλιστική, ε, ο θρηλυκός ε, Ολλανδικός ρεαλισμός, ο πραγματισμός πάρα πολύ επικοδομητικός σχετικά με την προσέγγιση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και το θέμα ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδέστηση, διότι η πρόοδη θα είναι άνισες. Μερικές χώρες θα προχωρήσουν περισσότερο πιο μακριά από τις άλλες χωρίς να κλείνουν την πόρτα στο σύνολο των 28 και βεβαίως το γεγονός ότι χρειάζεται ηγεσία, leadership πολιτικό ε, και ε, περισσότερες ε, γραφειοκρατικές δομές. Γάλλος είμαι, γι' αυτό υποστηρίζω αυτό το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ευστοχό. Εγώ βρήκα πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εάν μπορείς να μας δώσεις μερικές ενδείξεις σχετικά με τις, την, ανάπτυξη δυνάμεων από την Ολλανδία στο Μαλί, είναι μια πρόσφατη ε, απόφαση αυτή η δύναμη που θα αναπτυχθεί στο Μαλί. Έχω πολλούς συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Αρχίζουμε με τον κύριο Βαν Μπάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως είναι πολύ χαρά να βλέπουμε εδώ την Ζάνιν Χένες, πρώην συνάδελφο. Έχω ε, λίγες ερωτήσεις. Η Χένες είπε να μην γίνεται, ε, να μην υπάρχει επικάλυψη. Επικάλυψη δεν υπάρχει στρατός του ΝΑΤΟ, στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεργαζόμαστε καλά επί τόπου. Γιατί να μην στείλουμε μια τακτική ομάδα, ένα battle group στο Μάλι και νομίζω ότι αυτές θα είναι επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Δώσατε ένα παράδειγμα. Μερικοί λένε ότι ε, χρειάζεται κανείς ε, ένα στρατηγείο, μια δίκηση για το θέμα αυτό. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Ο κύριος Γκάλερ. Ε, αξιότιμε Υπουργέ, αξιότιμε συνάδελφε, σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για την σημαντική αυτή σύνοδο εδώ. Και συμφωνώ σε μεγαλύτερο βαθμό με την ανάλυση που κάνατε. Προσυπογράφω τα όσα είπατε. Θα πρέπει να φέρουμε το μερίδιο της ευθύνη μας. Θα πρέπει όντως να γίνουμε security provider, πάροχος ε, ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλήσατε επίσης πολύ σωστά για τις οικονομίες κλίμακας. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο, θα ήθελα όλοι να επιδείξουν ένα πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Θα ήθελα να βάλει ένα ερωτηματικό σε κάποια θέματα που αναφέρατε. Είπατε ότι δεν χρειαζόμαστε νέο στρατηγείο. Στις Βεξέλλες έχουμε όλα τα στοιχεία ενό ε, στρατηγείου. Έχουμε και ένα επιχειρησιακό κέντρο, δεν το ονομάζουμε επιχειρησιακό στρατηγείο, αλλά έχουμε όλα τα μεμονωμένα στοιχεία για τον προγραμματισμό. Μόνο η εφαρμογή, η εκτέλεση γίνεται από το εθνικό επίπεδο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσεγγίσουμε τη σκέψη αυτή προκειμένου να συλλέξουμε τα μεμονωμένα αυτά στοιχεία τα οποία ήδη υφίστανται και να τα συνενώσουμε σε ένα νέο στρατηγείο το οποίο δεν θα ήταν κάτι καινούριο. Θα είχε πολιτικό νόημα σε ό,τι αφορά το συντονισμό και την συνεργασία τώρα. Πολύ σωστά αναφέρεται ότι δεν πρέπει όλα να γίνονται με όλους και με τα 28 κράτη-μέλη, αλλά οι μικρότερες ομάδες έχουν νόημα μόνο όταν υπάρχει συντονισμός. Και αυτό νομίζω ότι θα αποτελούσε ένα καθήκον για την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, για να δώσει ακριβώς αυτή την επισκόπηση που έχετε για την συνεργασία. Γιατί μόνο από κάτω προς τα πάνω και συμμετοχή και των 28 κρατών μελών θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση καλύτερα να υπάρχει μια συντονιστική λειτουργία σε αυτό το επίπεδο που θα φροντίσει όσοι θέλουν να συνεργαστούν, να μπορούν να συνεργαστούν, να υπάρχει μια γενικότερη επισκόπηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα τρία envelopes, αυτοί οι τρεις τομείς, αυτοί οι τρεις φάκελοι που προβλέπονται στρατηγική, capacity, capability, ικανότητα και ό,τι αφορά την ιστορική αγορά, σε ό,τι αφορά την τυποποίηση και την πιστοποίηση. Αυτά τα τρία λοιπόν ζητήματα. Ποια? Ποιε είναι οι ελάχιστε προσδοκίε σα από τη Σύνοδο ό,τι αφορά του τρει τομεί αυτού. Και μια άλλη ερώτηση πολύ σημαντική και αυτή για τι αποφάσει τι οποίε θα χρειαστεί να πάρουμε εκ των υστέρων. Θα πρέπει να υπάρχει μία αναθεώρηση για θέματα άμυνας ένα stock taking, μια καταγραφή της κατάστασης για να δούμε τι θέλουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι χρειαζόμαστε. Μια αναθεώρηση λοιπόν για θέματα άμυνας μετά την ε, σύνοδο και τελευταίο σημείο για την ε, εκτέλεση των, αποφάσεων του Συμβουλίου. Μη ε, θα έπρεπε να τυποποιήσουμε, να δώσουμε ένα πιο επίσημο χαρακτήρα στις συναντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Άμυνας των Υπουργών Άμυνα για να μην συνεδριάζουν σε άτυπο επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Λίζεκ, ο αντιπρόεδρος Λίζεκ. Για να σας δείξω πόσο, ε, πόσο μεγάλη ποικιλία υπάρχει στο κοινοβουλίο μα θα μιλήσω πολωνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάρα πολλά άκουσα που με ενδιαφέραν ιδιαίτερως και αυτό με οδηγεί στις εξής δύο ερωτήσεις. Οι χώρε είναι μία από τις χώρες εκείνες που έχουν περικόψει τις ε, αμυντικές της δαπάνες. Οι σύμμαχοί μας δηλώνουν ότι οι περικοπές σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα. Θα μπορούσατε ίσως ε, και εσείς ε, να σχολιάσατε αυτή την εκτίμηση που την συμμερίζονται και πολλοί εμπειρογνώμονες. Δεύτερη ερώτηση, η Επιτροπός Ρέντινγκ πριν από κάποιες ημέρες δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δημιουργήσει τις δικές της ε, δυνάμεις, μια μυστική υπηρεσία ενδεχομένω. Ρωτώ λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ξεχωριστό τμήμα μυστικών ε, πληροφοριών. Yeah. Κύριος Στράσελ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμη Υπουργέ, αγαπητή Ζανίν. Χαίρομαι που σε βλέπω μετά από τόσο μεγάλη συνεργασία στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που στην Ολλανδία υπάρχει μια υπουργό άμυνα. Στην Γερμανία έχουμε και μια καγκελάριο η οποία ίσω να μην μα ικανοποιεί τόσο πολύ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί μιλώντας με τα στρατεύματα επιτόπου και με τις αμυντικές μονάδες διαπιστώνω ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με το τι γίνεται στην ε, Γερμανία στη σχετική πολιτική. Είπατε τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να γλιτώσουμε φορολογικές δαπάνες. Συμφωνώ και με τις περικοπές στα αμυντικά. Και αυτό ισχύει και για τη Γερμανία και για την ε, Ολλανδία, μιλώντας για το παράγωγο αυτό της ειρήνης είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πού θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας προκειμένου να γίνουν περαιτέρω περικοπές στην άμυνα. Γιατί και για τα θεωρηκτά και για τα στραταφέρματα ε, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη όπλων που είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά από την άλλη και σε ό,τι αφορά πολέμους εξ απόστασης. Εδώ λοιπόν οι απόψεις διήστανται. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη του Υπουργείου Άμυνης της ε, Ολλανδίας. Τι γίνεται και με τα μη επανδρομένα οχήματα. Ποια είναι δική σας άποψη. Είναι και αμφιλεγόμενο πολύ καθόλου το θέμα αυτό. Γιατί παράπλευρες ε, ζημιές που αποτελούν ε, μια φρικτή λέξη θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τους πολέμους εξ που διεξάγονται εξ Και αυτό δεν έχει να κάνει και πολλά πλέον, ξέρετε, με το πολεμικό δίκαιο στην παραδοσιακή του έννοια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάφ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που βλέπω την παλιά συνάδελφο που προήχθη ε, σε υπουργική θέση μεγάλης σημασίας. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στο σωστό μείγμα ε, στην παρουσία σας ανάμεσα στην απεσιοδοξία και στον πραγματισμό. Ε, δεν μπορούμε ε, να δεχθούμε, να παραδεχθούμε ότι τα δέκα τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει να κάνουμε σημαντικές πρόοδους προς την κατεύθυνση του σχηματισμού ε, μιας πολιτικής, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για την οποία θα μπορούμε να υπερεφανευόμεθα και αυτό δεν παρατηρήθηκε αλλού στον κόσμο. Συμφωνώ μαζί σας για να επιταχύνουμε το ρυθμό, για να έχουμε ένα αρχηγείο επιχειρησιακό ε, σε αυτό το σημείο είναι κάτι το πρόωρο. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε οι μεν τους δε στρατιωτικά προτού ασκήσουμε πίεση για ένα αρχηγείο, το οποίο θα πρέπει να είναι η κατάληξη. Το τέλος, συμφωνώ μαζί σας απολύτως ότι η συνεργασία πρέπει να σημαίνει συμμετοχή και ελπίζω ότι αυτό το δίδαγμα θα το μάθουμε εδώ, θα αντλήσουμε αυτό το δίδυγμα και θα το και θα το διαδώσουμε και στην Γερμανία που δεν κατάλαβε πάντοτε αυτό το μήνυμα, το ουσιαστικό μήνυμα. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αναφέρεται τις ε, επιδόσεις, επιδόσεις του Συμβουλίου Υπουργών όταν δρά ε, για την άμυνα, ως ε, υπεύθυνο για την άμυνα. Ε, πόσο αποτελεσματική ήταν η δράση του Συμβουλίου. Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο ε, το Συμβούλιο Υπουργών διαχειρίζεται τα θέματα άμυνας. Τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την εμπειρία ενώ πλησιάζουμε ε, ε, στην ημερομηνία διορισμού ενός διαδόχου της Κάθριν Άστον του χρόνου. Και το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται τον ε, την άποψη στρατηγικής στην άσφυλα και άμυνα που είναι μια στρατηγική που δεν είναι συντονισμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητηθεί μια κοινή λευκή βίβλος, αλλά λήψη αυτής πιστεύετε ότι ένα κοινό σχήμα, ένα κοινό πρόγραμμα για την εθνική, για τις αναφορές, για τις εκθέσεις εθνικής στρατηγικής δεν θα ήταν ένα κατάλληλο σημείο κίνησης για να προκαλέσουμε μεγαλύτερη συνοχή ε, και κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της παλαιάς συναδέλφου ως ε, Υπουργού Άμυνας αυτή τη φορά, να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου γιατί όλη την ενέργεια την οποία επέδειξε κατά τη διάρκεια της αιτίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αφιερώνει τώρα στην προώθηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ε, χαίρομαι για την προετοιμασία της Ολλανδικής Αποστολής στο Μαλί και πράγματι βρισκόμαστε σε μια φάση κατά τη διάρκεια της οποίας λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης τα κράτη-μέλη μειώνουν τους προϋπολογισμούς τους και βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μετακινούν το κέντρο βάρους της πολιτικής αμυνάς τους προς την Ασία και τον Ιεροϊνικό ωκεανό. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βελτιώσει και να αυξήσει και μάλιστα αρκετά σύντομα τις αμυντικές της ικανότητες και τις ικανότητες της στον τομέα της άμυνας και είδαμε, πήραμε κάποια πρώτα μαθήματα από την κρίση έτσι όπως εξελίχθηκε στη Λιβύη. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν πώς εκτιμάτε την συνεργασία μέχρι τώρα με τις Ηνωμένε Πολιτείες, πώς ακριβώς εκτιμάτε ακριβώς ε, την διατλαντική αυτή σχέση η οποία είναι κατεμένη γεγραμμένη στο ευρωπαϊκό DNA και σε ποιο βαθμό είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας ε, τις υποχρεώσεις μας στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας ε, και της, του ρόλου και της Τουρκίας. Ο κύριος Νταφ είπε ότι από τη μία έχουμε την δυνατότητα να είμαστε θετικοί, από την άλλη αρνητικοί και από την άλλη ρεαλιστές. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια διαφορετική ναυτικού τύπου θα έλεγα ορολογία Ε, νομίζω ότι ο αισιόδοξο περιμένει όπως λένε ο αισιόδοξο ναυτικός περιμένει να φυσήξει ο ούριος άνεμος, ο απεσιόδοξος θεωρεί ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά και ο πραγματιστής ναυτικός απλά ρυθμίζει τα πανιά του για να προχωρήσει το ταξίδι του. Ευχαριστώ κυρία Σάκα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Βεβαίω θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την πρώην συνάδελφό μα που έγινε υπουργό. Δύο ερωτήσει διότι πάρα πολλά λέχθηκαν. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή σας θεώρηση για σχετικά με την ευρωπαϊκή άμενα σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο είναι πάρα πολύ εύστοχη κυρίως εφόσον έχουμε έλλειψη δυνατοτήτων και πολιτικής βούλησης, κυρίως όσον αφορά στη Συρία. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα σε σχέση με το θέμα αυτό, σε συνδυασμό με την διπλωματία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Τι επιλογές έχει η Ευρώπη, υπάρχουν στρατιωτικές επιλογές ή πώς αλλιώς μπορούμε να επιδείξουμε ένα leadership, ένα ηγετικό ανάστημα στο θέμα αυτό. Βεβαίω, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο κανεί να έχει αυξημένη, ενισχυμένη συνεργασία όταν υπάρχουν ριζωμένα συμφέροντα σε νέου τομείς ε, Άμυνα, όπως τον κυβερνοχώρο. Είναι, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κανόνες εξ αρχή η συνεργασία εξ αρχής. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σα, όταν, όταν πρόκειται για νέου τομεί άμυνα. Υπάρχουν νέε επιλογέ Ευρωπαϊκή συνεργασίας ευθύ εξ αρχή, Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Υπουργέ, σας δίνω τον λόγο. Πολλοί συνάδελφοι, πολλές ερωτήσεις. Ίσως η ιδιαίτερη διάταξη της αίθουσα αυτής ε, να σας ε, προβληματίζει, διότι περιμένουμε και συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά έχουμε την ποιότητα των ερωτήσεων που δείχνει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η η ε, παρουσία σας. Αν μου το επιτρέπετε θα συνεχίσω στα Ολλανδικά διότι θέσατε πολλές ερωτήσεις και είναι ευκολότερο για μένα. Σε ό,τι αφορά το νέο αρχηγείο, το νέο headquarters, το νέο στρατηγείο, πολύ καλά είπε ο κύριος Νομίζω ότι ε, αν ξεκινήσει η συζήτηση γι' αυτό θα χάσουμε την ουσία. Φυσικά υπάρχει το επιχειρησιακό κέντρο, αυτό το αρνούμε και αυτό έχει σημασία, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από μια κεντρική γραμμή ε, συντονισμού από ένα κεντρικό στρατηγείο. Αυτό οργανώνεται και διοργανώνεται αναποστολή. Αυτό το μπορούν να το επηρεάσουν και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ε, ικανότητες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το, αυτό και αυτό το επενούμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε Ίσως σε τελική ανάλυση αυτό προκύψει. Αλλά η Ευρώπη γενικά είναι μια μακριά, μακρόπνοη διαδικασία. Ας βελτιώσουμε λοιπόν τώρα την ε, συνεργασία και την ενσωμάτωση όλων αυτών των μονάδων. Καταλαβαίνω τι λέτε βέβαια. Ρωτήσατε και για θέματα εσωτερικής ε, αγοράς. Ανησυχώ γι' αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορα συμφέροντα από τις ε, διάφορες χώρες. Να μην το αρνούμαστε αυτό. Για μας, για την Ολλανδία, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τους ε, υπανάδοχους, τους υπεργολάβους, τις μικρές αυτές επιχειρήσεις, οι οποίοι στη μεγάλη συζήτηση αυτή ίσως ε, να μην τους δίδεται η απαραίτητη προσοχή, το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Το συζήτησα και με τους επιτρόπους. Θα συνεχίσουν να το θέτω το θέμα αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε σε τελική ανάλυση όλα τα κρατημέλη να έχουν επισκόπηση πέρα από τα σύνορά τους και να μην δρούν μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ρωτήσατε επίσης ποιος είναι ο ρόλος της ΕΝΤΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που δραματίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνης. Ε, έχουν ε, επαρκεί μέσα για να δραματίζουν το ρόλο του στην παρούσα φάση. Και αυτό το είπε πάρα πολλά η κυρία Σχάκε. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και στα κρατημέλη. Η έκκληση της ΕΝΤΑ για πιο πολλά χρήματα, πιο πολλή κονδύλια, θεωρώ ότι πάντα αποτελεί ένα πρόβλημα, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περικοπές, αντιμετωπίζουν μεσογενικά προβλήματα και αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα, οι δαπάνε αυτές είναι απαραίτητες και ότι πραγματικά συνδράμουν ε, στην ε, ενίσχυση των κρατών μελών. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε φυσικά και στα μέσα Νοεμβρίου. Ο κύριος Λίζεκ. Ρωτήσατε και είπατε ότι η Ολλανδία έκανε σημαντικές περικοπές στην άμυνα όπως και άλλα κρατημέλη. Όντως, αυτό στέκει. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει η ειρήνη. Μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου έγιναν τεράστιες αναδιοργανώσεις. Και δεν μπορώ να αρνηθώ ότι και προσφάτως έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές. Αλλά σε κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι κοιτάξτε αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πράξη. Αλλά στην πράξη πολλοί ε, κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί χρειάζονται αυτές οι δαπάνες, γιατί θεωρούν ότι αυτή η ασφάλεια ειρήνη που επικρατεί στην ε, Ολλανδία, στην οποία και μεγάλωσα, ε, δεν βλέπουν ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προασπιστούμε απαραίτητα για τη δική μας εμερία, για τη δική μας ε, ειρήνη και πέρα από τα σύνορά μας. Χρειαζόμαστε ψηλή ποιότητα σε τέτοια θέματα. Και αν με ρωτήσετε λοιπόν ε, κατά πόσον έχω φιλοδοξία, κατά πόσον θέλω και άλλε δαπάνε, ναι, βεβαίω, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικονομική πραγματικότητα. Αλλά να σας ε, διαβεβαιώσω ότι στην Ολλανδία μπορούμε να συνδράμουμε στο παγκόσμιο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τα στρατεύματα, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπερμαχός, μίλησατε για τις μάχημες ομάδες, τις ομάδες μάχης και για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή το σύστημα αυτό. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ω τώρα, αλλά σας είπα, ή θα τα χρησιμοποιήσουμε ή θα τα χάσουμε αυτά ως δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό το είπα και στην αρχική μου παρέμβαση να δείξουμε και για τις ε, ασκήσεις και για να τα επιδείξουμε τα στρατεύματα μας ε, για το Ευρωπαϊκό στρατό, για το στρατό του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι υπέρμαχος και πιστεύω και εμένω σε αυτό. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που τελικά ε, θα πρέπει να καθορίζουν κατά πόσον θα επιστρατεύσουν, κατά πόσον θα αναπτύξουν τις δυνάμεις τους. Φυσικά χρειάζεται μια κεντρική καθοδήγηση για τον συντονισμό των στρατευμάτων, αναμφίβολα ο κύριος Φαμπάλε ρώτησε. Συγγνώμη να βρω την ερώτηση του κυρίου Φαμπάλε. Ρώτησε τι ισχύει για τις ε, ομάδες ε, μάχης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα battle groups. Ναι, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για το force protection. Γιατί όχι. Αν δημιουργηθούν τέτοιες δυνατότητες, γιατί να μην καλυφθούν τρει, τρεις-τέσσερις ε, πρώτοι μήνες προκειμένου και σε ό,τι αφορά θέματα δημιουργίας τέτοιων δυνάμεων να δοθεί κάποια ανάσα. Νομίζω ότι για τις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, σύμφωνοι, ναι, δεν υπάρχει κάποια στάνταρ ε, ε, συνταγή. Πάντα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την, την πιθανότητα κλιμάκωσης. Ποτέ δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση. Για τα... το αρχηγείο το οποίο θα πρέπει να έχει πλήρες δυναμικό. απάντηση σε αυτή την ερώτηση για να μην ε, πλατιάσουμε σε μια θεωρητική κυρίως συζήτηση, να παραμείνουμε με τα δύο πόδια όπως λέμε ε, στο έδαφος ρεαλιστές, να δούμε τι ισχύει στην πράξη και τι χρειαζόμαστε στην πράξη. Ρωτήσατε επίσης ε, για το τι μας αποδίδει η ειρήνη. Νομίζω ότι αυτό το απολαμβάνουμε ήδη. Πολλές περικοπές έχουν γίνει στην Ολλανδία και σε κάποιες, ε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει ε, αν θέλετε, στο απόλυτο ελάχιστο, αλλά θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τα ελλανδικά στρατεύματα είναι υψηλή ποιότητα για τι ε, δυνατότητε συνεργασία Wolfgang. Είναι απεριόριστε. Ε, μίλησα με τον κύριο Τόμα Μαζέρε, τον Γερμανό Υπουργό. με επιστολή προθέσεων σε ό,τι αφορά συνεργασία Γερμανία και Ολλανδία, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη συνεργασία των αέριων μονάδων μας εξετάζουμε δυνατότητες υποβροχίων και κοινή εκμετάλλευση. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό μπορούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν δυνατότητε τι οποίε πλέον μόνε του οι χώρε δεν μπορούν να αναπτύξουν. Ανέφερα τη Γερμανία, αλλά και την Πολωνία και την Πολωνία που πάλι συνεργάζεται με την Ολλανδία. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται μικρές ομάδες κρατών που συμμετέχουν σε τέτοιες συνεργασίες. Άρα λοιπόν για τις δυνατότητες συνεργασίες σε καμία περίπτωση δεν τις έχουμε εξαντλήσει. Ο κύριος Άντριου Ντάφε μίλησε πολύ σοφά με τα για το επιχειρησιακό αρχηγείο, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Να σχολιάσω την ε, Λέδη Άστον μου ζήτησε επίσης δημοσίως. Νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή να γίνει μια έκθεση αξιολόγησης. Ε, αλλά όπως είπε η κυρία Σχάκε, το θέμα είναι η πολιτική βούληση, η πολιτική βούληση 28 κρατών μελών. Και φυσικά υπάρχει η Λαδιά δηλαδή, φυσικά και υπάρχει ο κύριος Μαρόμπαϊ, οι οποίοι επίσης πρέπει να κληθούν και να επιδείξουν πολιτική βούληση, πολιτική δέσμευση. Αλλά αυτό ισχύει και για τα 28 κράτη-μέλη, γιατί δεν πρέπει στο Συμβούλιο να φτάνουμε και να βλέπουμε ένα τείχος απροσπέλαστο τελικά. Θα πρέπει να διδραματίσουν και οι Λεδιά και ο κύριος Μαρόμ πάει το ρόλο τους, αλλά θα πρέπει και τα 28 κρατημέλη να σημειώσουν πρόοδο. Μιλήσατε για ένα common template. Νομίζω ότι αναφέρεστε κυρίως στα σχέδια δυνατοτήτων, ικανοτήτων και ναι, πρέπει να πω ότι αυτά θα πρέπει να τα μοιράζονται τα κράτη-μέλη, γιατί μόνο τότε υπάρχει το Military Short Force και αν υπάρχουν αυτά τα σχέδια λοιπόν ικανοτήτων μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να καλύψει τι, πού υπάρχουν κενά, πώς μπορούν να πληρωθούν τα κενά αυτά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό από κοινού. Αυτό είναι πολύ καλό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούμε όλοι να αγοράζουμε ε, και να μην έχουμε τελικά ελικόπτερα. Όχι. Θα πρέπει κοινά να γίνονται αυτές οι επενδύσεις. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί και την ουσία της έκθεσης της κυρίας, της δηλαδή Άστον. Ο κύριος Σαραφράγκα μίλησε για τις περικοπές. Το είπα είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και αυτό έχει αντίκτυπο και στις ε, δαπάνες, στις αμυντικές. Ποτέ όμως σε καμία περίπτωση δεν θα διακυβεύσουμε την ασφάλειά μας, την ειρήνη μας. Δεν είναι πράγματα αυτονόητα, ποτέ δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε αυτονόητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις. Αυτό το ζητώ από τον εαυτό μου ως Υπουργό Άμυνας, από τους άλλους Υπουργούς Αμήνης, από εσάς. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να ενημερώνουμε το ευρύ κοινό. Γιατί συχνά ξέρετε ο κόσμος έχει μεν μεγάλο σεβασμό τρέφει προς τους στρατιωτικούς στο στρατό, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί γίνονται αυτές οι δαπάνες. Γι' αυτό λοιπόν όλοι θα πρέπει να αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας και όλοι θα πρέπει να αισθανόμαστε την ευθύνη για την... Ε, για τις είπα, εξαιρετικός εταίρος για την Ευρώπη και θα παραμείνει εξαιρετικός εταίρος, αλλά κανείς νομίζω δεν ε, αγνοεί το γεγονός ότι γίνεται μια τεράστια συζήτηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για την επιμερισμό των ευθυνών. Burden sharing. Οι ΙΠΑ την ευθύνη τους, η Ευρώπη ε, είναι ακόμα κατακαιρματισμένη. Αυτή τη συζήτηση λοιπόν την διεξάγουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον για να είμαστε πιστικός πάροχος ειρήνης, αξιότιμος ομόλογος των Ιπα. Οι Αμερικάνοι λοιπόν θέλουν πραγματικά να δοθεί νέα πνοή και νέα μορφή στην συνεργασία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ μπορεί να μας ωφελήσει. Μπορεί αυτή η διαθελοντική συνεργασία είναι σημαντική, θα παραμείνει σημαντική. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να ζητήσουμε διακοπή αυτής. Νομίζω αρκετά είπαμε για τη Λέδη Άστον και για τον κύριο Φαρόμπα για την πολιτική βούληση της Μαρία Ντεσχάκερ. Τα ανέφερα αυτά επαρκώς θεωρώ όταν έπτυξα. Ναι, και με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί τελικά πρόκειται για μια κοινή πορεία. Αυτή η ο διαφορετικό διάλογος έχει σημασία. Η συνεκτική προσέγγιση, ε, αυτό το στοιχείο, τα τρία στοιχεία της προσέγγισης, και τα βλέπουμε αυτά και στο Μάλι και στη Συρία όπου όμω είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία με τα χημικά όπλα για σουτέις, λέει η κυρία Ένες Πλάσκαρτ. Έχουμε λοιπόν μια νέα κατάσταση. Ε, είναι επικίνδυνο θεωρώ να σχολιάσουμε στην παρούσα φάση. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση μια στρατηγική παρέμβαση δεν θα οδηγήσει πουθενά αλλά πιστέψτε μα ότι σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην κορυφή του πρωτοβουλίου μας το θέμα αυτό για το Μάλι τώρα. Η Ολλανδία αποφάσισε να συνεισφέρει σημαντικά. Έχουμε και το EUTM. Θα συνεισφέρουμε δυνάμεις στη Μιουνίσμα την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν και περαιτέρω δυνατότητε συμβολής. Όλοι φυσικά παραπονιόμαστε ε, για το λαθρεμπόριο ανθρώπων, ε, όπλων, ναρκωτικών, την ε, παράνομες ροές μεταναστών, την πίεση στα εξωτερικά μας σύνορα. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη χώρα προέλευση, στη χώρα διαμετακόμισης, να μην περιμένουμε να μας χτυπάν την πόρτα, να μας χτυπάν στα σύνορά μας τα προβλήματα. Αυτά. Πρόεδρο, νομίζω απάντησα σε όσε πιο πολλέ ερωτήσει μπορούσα. Συνεχίζει η κυρία ε, Πλάσχαρτ. Ε, Μιλάτε τέλεια ε, Ολλανδικά. Ρωτήσατε όμω, κύριε Γκάλερ για το άτυπο συμβούλιο. Θέλετε να δοθεί ένα επίσημο χαρακτήρα στο άτυπο αυτό συμβούλιο. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Είναι λίγο θεσμικό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαι υπέρμαχος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Νομίζω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Ευχαριστώ άλλη μια φορά που ήρθατε κατόπιν δικής μας προσκλήσεως. Ελπίζω ότι μετά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια για την έναρξη μιας διαδικασίας. Είσαστε πάντοτε πρόσδεκτοι Ξέρετε πολύ καλά το χώρο και θα είναι μεγάλη χαρά να σας ξαναβρούμε εδώ ή στα πλαίσια της ΑΦΕΤΑ Ευχαριστώ άλλη μια φορά στην συμμετοχή της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Θα διακόψουμε για λίγη ώρα. Ευχαριστώ σε εσά και ε, σας εύχομαι ε, καλό κουράγιο. Liebe Kollegen, sehr geehrte Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ως ε, ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, χαίρομαι που μπορώ να σα καλωσορίσω εδώ σήμερα. Δυστυχώ ο πρόεδρο μα ε, είναι άρρωστο ο Χέρμαν Μπρόκ, και αυτό μου ζήτησε να προεδρεύσω. Το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Πολιτική άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη τη Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία που θα συμπεριλαμβάνει συζήτηση και με εσά, εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων, που παίζετε σημαντικό ρόλο. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι η παρουσία σα εδώ και οι παρεμβάσει σα θα είναι σημαντικέ για τη δημιουργία μια συνεκτική πολιτική άμυνα. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας και εξηγώντα του λόγου για του οποίου είναι σημαντική η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα σε ό,τι αφορά τι προσδοκίε και τι ελπίδε των Ευρωπαίων και σε ό,τι αφορά και την μετεξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όποιο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζούμε, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν όλοι για το πώς αλλάζει ο κόσμος και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε στο μέλλον σε θέματα ειρήνης κυρίως. Και υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα οποία επιδρούν και στην καθημερινή ζωή των πολιτών στην Ανατολή, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διαρκώς ε, ε, δοκιμάζει τις δυνάμεις της και τους μίστης, αν θέλετε, η Ρωσία, καταπιέζοντας τους γείτονε Ανατολά. Στον ε, Νότο έχουμε την Αραβική Άνοιξη και τις ε, τριβές μεταξύ των ε, ριζοσπαστικών Ισλαμιστικών δυνάμεων και των επαναστατικών δυνάμεων. Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από εμά τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά να εγγυηθούμε τα πρότυπα και το επίπεδο ζωής και τις ελευθερίες τους, να εγγυηθούμε το μέλλον τους. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική χρειάζεται μια νέα δυναμική που θα βασίζεται στις καινοτομίε της ε, συνθήκης της Λισαβόνας που μας επιτρέπουν να σημειώσουμε οικονομική και κοινωνική πρόοδο προασπίζοντας τις αξίες και τα συμφέροντά μας σε όλο τον πλανήτη για να μπορέσουμε να δώσουμε ενίσχυση ε, στην κοινή πολιτική μας και να βελτιώσουμε τις ε, δυνατότητες ε, άμυνας, χρειαζόμαστε πιο πολύ συνοχή και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αλλά όλος ο ιδιαίτερος χρειάζεται να υπάρχει αξιόπιστες δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας προκειμένου να αποφύγουμε συγκρούσεις, να ανταποκριθούμε σε συγκρούσεις και να μπορέσουμε να προασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι τόσο σημαντικά. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής. Εδώ και 25 χρόνια σχεδόν από το τέλος του ψυχρού πολέμου θέλουμε να μειώσουμε τις ε, αμυντικές περικοπές και τις μειώνουμε. Όλος παραδόξως, ο αριθμός των επιχειρήσεων όμως στις οποίες εμπλέκονται τα ευρωπαϊκά στρατεύματα έχει αυξηθεί και μάλιστα κατά πολύ. Αυτό τι σημαίνει ότι οι επενδύσεις στα αμυντικά και στους εξοπλισμούς ε, είναι πτωτικές, πτωτικής τάσης, αλλά η ζήτηση αυξάνεται και αυτή η τάση μας ενοχλεί εδώ και πολύ καιρό. Πολλούς εξημώνει, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι οι στρατιώτες μας, εν ώψη και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν εξ ονόματος όλων των Ευρωπαίων, χρειάζονται την πλήρη μας υποστήριξη. Και επιπλέον, η, ευρωπαϊκή, η παγκόσμια κρίση, η οικονομική κρίση, σημαίνει και περτέρω περικοπή σε ανησυχητικό επίπεδο των αμυντικών δαπανών. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερως είναι ότι οι περικοπές αυτές γίνεται με πλήρως ασυντόνιστο τρόπο. Ναι, υπάρχουν κάποιες μεν ε, διμερείς και αν θέλετε και τριμερείς, τετραμερείς ε, συζητήσεις και συντονισμοί, αλλά σε γενικές γραμμές το ευρύτερο σύνολο χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισμού. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι επικίνδυνη, αλλά και περιττή. Επικίνδυνη γιατί το παγκόσμιο προσκήνιο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και θα ξεκολουθήσουμε να χρειαζόμαστε κάποιες αμυντικές δυνατότητες. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας έχει δώσει τα εργαλεία για ένα καλύτερο συντονισμό και για την ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων. Θέλουμε το πλαίσιο λοιπόν αυτό της συνθήκη της Λισαβόνας να το εξαντλήσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε έναν ευρωπαϊκό συντονισμό προκειμένου να μην χάσουμε πιο πολλά κρίσιμα συστατικά της ε, πολιτικής μας, για τους ε, στρατηγικούς μας στόχους, για τις στρατηγικές μας επικοινωνίες, ε, τους δορυφόρους, τις δυνατότητες ανεφοδιασμού στον αέρα. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο. Αλλά ε, επιτρέψτε μου να επισημάνω δύο-τρία συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία απαραίτητο θα πρέπει να συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να καταστρωθεί ένα οδικό χάρτη με σαφέ χρονοδιάγραμμα για ει βάθο συντονισμό στον τομέα τη άμυνα. Η εφαρμογή δε μιας μόνιμης διαρθρωτικής συνεργασίας ενός συνασπισμού των προθύμων θα πρέπει να προωθηθεί ενό τέτοιου πυρήνα. Και αυτό θα πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και θα πρέπει να υποστηριχθεί η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά όλες αυτές οι ιδέες θα ωφελήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πεπισμένος ε, προασπιστής της ε, συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των διακρατικών σχέσεων, αλλά και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ιδίων μας ικανοτήτων να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι είμαι απογοητευμένος γιατί κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί μας δήλωσαν ότι το Δεκέμβριο δεν θα πρέπει να επιτύξουμε τόσο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία, γιατί το ευρωπαϊκό κοινό δεν είναι υπέρ μια τέτοια συντονισμένη στρατιωτική ανάπτυξη. Φυσικά δεν το απασχολούν το κοινό τεχνικέ λεπτομέρειε. Παρ' όλα αυτά όμω οι πολιτικοί θα πρέπει να ασχοληθούν με τέτοια θέματα αυτά για να εξεύρουν λύσει που θα καθησυχάσουν τις ανησυχίες των πολιτών μας. Απογοητεύομαι επίσης, γιατί δεν πιστεύω πραγματικά ότι οι Ευρωπαίοι δεν νοιάζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική και για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όταν μιλώ με τους Ευρωπαίους για τις προσδοκίες και για τις ανησυχίες τους, διαπιστώνουμε ότι τις ανησυχεί η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές που σημαίνει αυτές, ε, αυτή και ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή και ξέρουν ότι κοστίζει πολύ όταν ξεσπάει μια σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνονται οι τιμές των υπολογιστών, γιατί αυξάνονται τιμές ε, στις, ε, στα ορεκτά η Κίνα και ότι κινδυνεύει η υγεία των παιδιών τους όταν σημειώνονται προβλήματα στις κοντινές μας περιοχές. Σε ό,τι αφορά και τις ροές μεταναστών, πρέπει να διευκρινίσω ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά πράγματα ως Ευρώπη για την επίλυση των διαμαχών επιτόπου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν συζητούμε καθημερινά τέτοια ζητήματα και βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συνεργασία για να ανταποκριθούμε σε αυτή την μεταβαλλόμενη παγκόσμια κατάσταση και το ξέρουμε ότι οι πολίτες μας είναι πιο ε, συνειδητοποιημένοι από ό,τι θεωρείται όταν λοιπόν συνερχόμαστε κάθε έξι μήνες με τα εθνικά κοινοβούλια ξέρουμε ότι θα ακούσουμε και ότι θα έχουμε παρόμοιες απόψεις, οπτικές γωνίες μαζί με εσά μπορούμε να, να εισακουστούμε από τους Ευρωπαίους πολίτες να διασφαλίσουμε ότι στην πολιτική την εξωτερική μας και την πολιτική της άμυνας μπορούμε να σημειώσουμε πραγματικό αντικτύπο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πραγματικά θα πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τις ευθύνες τους και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκέμβριου θα πρέπει να λάβουν σημαντικές απαντήσεις, αποφάσεις. Θα πρέπει να δράσουν για να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων, των διεθνών περιστάσεων και μάλιστα αν θέλουν να έχουν κάποια επιρροή στις μεταβολές, στις αλλαγές αυτές του παγκόσμιου προσκυνείου. Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση με τους εκπροσώπους των 28 κρατών μελών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, τον κύριο Ντανζόν. Ευχαριστώ, Αντρέη. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας καλωσορίζω εδώ στο ημικύκλιο ο κύριος Κοβάτσεφ παρουσίασε την κατάσταση, θα ήθελα απλώς ως εισαγωγή να σα υπενθυμίσω ότι τελικά το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το ερώτημα που θέτουν οι συμπολίτες μας και επαναλαμβάνω τα όσα λέχθηκαν στην εισαγωγή. Δεν νομίζω ότι οι συμπολίτες μας δεν ενδιαφέρονται για την άμυνα και την ασφάλεια και έχουμε κρίσεις που πολλαπλασιάζονται στο περιβάλλον μας και το ακούτε, ακούτε τι απασχολεί τους συμπολίτες σας στις εκλογικές σας περιφέρειες ε, το θέμα που ακούμε για το Μαλή, για τη Συρία, για τη Λιβύη είναι τι κάνει η Ευρώπη, πού βρίσκεται η Ευρώπη στα θέματα αυτά. Υπάρχει ε, ερωτήματα που τίθενται σχετικά με την θέση που θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη στην διεθνή σκηνή, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη. Τα ευρωπαϊκά όργανα είναι ακόμα νέα ως προς τον τομέα αυτό. Είναι εντογίγνεσθε, υπάρχουν, αλλά η πρωταρχική πολιτική ευθύνη ανήκει στα κράτη-μέλη. Και εσείς παίζετε έναν κρίσιμο ρόλο και είναι απαραίτητο να έχουμε μια διαβούλευση, συνεννόηση αρκετά στενή για να προωθήσουμε αυτό το θέμα, αυτή την υπόθεση που ενδιαφέρει ε, τους συμπολίτες μας ε, και που είναι νόμιμη λόγω της εξέλιξης ε, του στρατηγικού πλαισίου που υπενθύμησε ο Αντρέη Κοβατσέφ. Αν μου το επιτρέπετε, θα ήθελα απλώς να σας καλέσω ως Εθνικά Κοινοβούλια να επιμείνετε μαζί μας πριν από αυτό το Συμβούλιο πάνω στην χρησιμοποίηση, στην προώθηση αυτού του οποίου, το οποίο ήδη υπάρχει, διότι είμαστε πάρα πολλοί που πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αν είναι μια σημαντική ευκαιρία, δεν θα καταλήξει οπωσδήποτε σε θεαματικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, αλλά πάντως το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι τελείως ανύπαρκτη στον τομέα αυτό. Υπάρχουν μέσα, υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν αποστολές, υπάρχουν επιχειρήσεις που διεξάγονται κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άποψη αυτή και ήρθα από το Αφγανιστάν όπου πήγα την περασμένη εβδομάδα όπου υπάρχει μια αποστολή αστυνομική περίπου 400 ατόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα τα εθνικά κοινοβούλια να αποδώσουν λίγο περισσότερη σημασία σε αυτές τις αποστολές και επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν γνωρίζουν πολύ καλά οι συμπολίτες μας αλλά ακόμα και οι εθνικοί βουλευτές να επισκεφθείτε αυτές τις αποστολές, αυτές τις επιχειρήσεις, να καλέσετε τους επικεφαλείς των αποστολών σε ακροάσεις στα εθνικά σας κοινοβούλια. Μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα για το τι λειτουργεί καλά, για το τι λειτουργεί λιγότερο καλά και για το τι δεν λειτουργεί καθόλου. Αλλά με βάση αυτές τις ε, διαπιστώσεις θα μπορέσουμε να ελπίσουμε μία πρόοδο σε όλο το μηχανισμό τον ευρωπαϊκό, ο οποίος είναι ακόμα πάρα πολύ νέος ε, προς την πολιτική ασφάλειας ε, και άμυνας. Και ακούω τις διαπιστώσεις στα κράτη-μέλη μας. Πού βρίσκεται η Ευρώπη, τι κάνει η Ευρώπη, αλλά η πρωταρχική ευθύνη ανήκει στα κρατη και δεύτερον όταν η Ευρώπη κάνει κάτι θα πρέπει να ξέρουμε, να το αναγνωρίσουμε και ε, να το εκφιάζουμε, να το ε, προβάλλουμε. Αυτό βεβαίως δεν μας απαλλάσσει από το να ασκήσουμε τις ευθύνες μας επίσης και να είμαστε φιλόδοξοι. Από την άποψη αυτή θα πρέπει η ατζέντα, η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου αυτού να είναι αρκετά καλή. Έχουμε ε, τρία πράγματα, την ορατότητα, τις δυνατότητες, την βιομηχανική πολιτική. Τα τρία αυτά σημεία θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα σε αυτό το Συμβούλιο και θα πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη ούτως ώστε να ασχοληθούν με την καρδιά του θέματος και όχι απλώς να τα εξετάσουν επιφανειακά τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα ακούσουμε τον Ματσέλ Ποκοφσκή από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, που ασχολείται με την αμάνια και κοινή ασφάλεια και άμυνα και μετά από τον κύριο Ποπόφσκη προτείνω να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συνάντηση σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία για μας διότι τη θεωρώ ως μέρος της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για το Δεκέμβριο. Δεν είναι μόνο διακυβερνητική διαδικασία, βεβαίως κάνουμε πολλή δουλειά με τα κράτη-μέλη, αλλά είμαστε ευγνώμονες για αυτήν την ευκαιρία, διότι θα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Το θέμα της κυριαρχίας τίθεται εδώ και είναι σημαντικό και έχουμε περιορισμούς από ε, το θέμα της κυριαρχίας στη συζήτηση και είναι σημαντικό να έχουμε την πλήρη υποστήριξη του, των κοινοβουλίων. Κατά κάποιο τρόπο το 2013 ήταν ε, μια, ένα, μια, ένα έτος όπου αποδόθηκε πολύ σημασία στην ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει την ασφάλεια και την άμυνα δημιούργησε πολλές προσδοκίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλά άλλαξε επίσης ε, και το πνεύμα της συζήτησης στην στάση ε, που έγινε πολύ πιο θετική από ό,τι στο παρελθόν. Γνωρίζετε πολύ καλά την εργασία που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έκθεση της κυρίας Κοπά, του κυρίου Γκάλερ και τις εκθέσεις ε, τις μελλοντικέ του κυρίου Μπρόκ από, ξέρετε τι έχει γίνει από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, την Επιτροπή και το, την έκθεση που έκανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπα τη εκπρόσωπος. Ε, στις 11 Οκτωβρίου είχαμε την τελική εκδοχή και είχαμε ανταλλαγές με το Κοινοβούλιο και ξέρετε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά για την αγορά και την βιομηχανία άμυνας που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο και καλύψαμε νομίζω ένα μεγάλο μέρος του θέματος και είχαμε ε, επίσης από, τις, ε, από πανεπιστημιακούς φορείς, από την βιομηχανία είχαμε συμμετοχές, συνεισφορές που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για την τελική έκθεση της ΕΠΑ εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να σας πω ποια είναι τα επόμενα βήματα και να πω κάτι για την διαδικασία παρακολούθησης μετά το Δεκέμβριο για τα μελλοντικά βήματα. Δεν πρόκειται να συνοψίσω την έκθεση για σας, είναι διαθέσιμη, είναι ουσιαστική και το feedback που λάβαμε μέχρι τώρα τις αντιδράσεις των κρατών μελών αλλά και επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΝΑΤΟ ήταν μια αντίδραση θετική και ενθαρρυντική. Η έκθεση αρχίζει με μια σύντομη ανάλυση ε, του μεταβαλλόμενου γεωστρατηγικού πλαισίου, ε, τας προκλήσεις, ε, την μείωση των προϋπολογισμών των εθνικών που ανέφερε ο Πρόεδρος και από την άλλη πλευρά ως Ευρώπη αυξανόμεθα στον ε, κόσμο των παραχαίων άμυνας. Χρειάζεται λοιπόν μια στρατηγική συζήτηση για το μέγεθος της φιλοδοξίας μας ε, και για το πολιτικό επίπεδο. Η έκθεση ε, περιλαμβάνει τρεις συνεργατικούς σχηματισμούς, ορατότητα, δυνατότητας και τεχνολογική και βιομηχανική βάση, αλλά υπάρχει ήδη εδώ μια επεξήγηση, βλέπουμε τι πρέπει να κάνει η Ένωση για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και να προβάλλει τις αξίες της. Θα πρέπει να μπορούμε να δράσουμε διαμέσου της ΚΠΑΑ ως παροχέας, αλλά αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι χρειαζόμαστε δυνατότητες, ικανότητες και δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη. Και καινοτόμο βιο, ε, βιομηχανική βάση για να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Βεβαίως πρόκληση είναι πώς θα επικοινωνήσουμε με το κοινό μας και είναι εδώ μια ευκαιρία για τους ηγέτες θα είναι να διατυπώσουν μια επιχειρηματολογία θετική και να πείσουν ε, το κοινό ότι η άμυνα δεν είναι πολυτέλεια ούτε όχληση. Είναι κάτι που θα πρέπει ε, να επιδιώκουμε και που απαιτεί ε, δεσμεύσεις και επενδύσεις, όχι μόνο χρηματικές αλλά και άλλες. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες όταν θα συναντηθούν το Δεκέμβριο θα πρέπει να δουν ποια είναι η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη και των δυνατοτήτων και για το θέμα της μείωσης των δαπανών στα κράτη-μέλη. Και είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επισημάνει ορισμένες ευκαιρίες και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε το, ε, τις δυνητικές ε, δυνατότητες που έχουμε, που καμιά φορά υποτιμώνται, αλλά έχουμε και μια βιομηχανία με 100 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ατησίως ε, για και που δημιουργεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. 5.000. Η έκθεση της ΥΠΑ της εκπροσώπου αναφέρεται με το θέμα που συζητήθηκε δημόσια τα τελευταία χρόνια που το θέμα του ναι ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα στρατηγική ασφαλείας. Και μπορώ να αναφέρω από το ίδιο το κείμενο που λέει ότι ως μέρος της παρακολούθησης μετά το Δεκέμβριο τα κράτη-μέλη το επιθυμούν μπορεί να αρχίσει ευρωπαικη ενωση χρειαζεται μια νεα στρατηγικη ασφαλειας και μπορω να αναφερω απο το ιδιο το κειμενο που λεει οτι ως μερος της παρακολουθησης μετα το δεκεμβριο τα κρατη μελη το επιθυμουν μπορει να αρχισει εργασια για να προσδιοριστεί η στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης μέσα στον μεταβαλλόμενο πλαίσιο μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ μιας λευκής βίβλου ή μιας νέας στρατηγικής. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία το όνομα, αλλά η διαδικασία της, ε, του στρατηγικού προβληματισμού. Βέβαια, είπατε εκπρόσωπος δεν ήθελε να προκαταλάβει το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελε να αρχίσει αυτή η άσκηση αν τα κράτη-μέλη το Τώρα τι θα συμβεί μετά. Ανέφερα μερικές προπαρασκευαστικές ε, συζητήσεις στο Συμβούλιο, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας θα αφιερώσουν πολύ προσοχή στην ασφάλεια και άμυνα στις 18 και 19 Νοεμβρίου ε, με η οποία θα προηγηθεί της 13ης Νοεμβρίου του Συμβουλίου Ενέργειας, του Ενεργειακού Συμβουλίου που θα συναντηθεί στις 19 Νοεμβρίου επίσης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει πορίσματα που θα καλύψουν ε, τους τρεις συνεργατικούς συχηματισμούς που ανέφερα, τις τρεις ομάδες, αλλά είναι μια ευκαιρία για τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων να συζητήσουν, όχι μόνο να υιοθετήσουν πορίσματα, να συζητήσουν τα επίμαχα θέματα η εργασία άρχισε και ε, για το υπουργικό, την υπουργική συζήτηση και τη συζήτηση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος, διότι ξέρουμε ότι ο βαθμός επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι περίπου 50% σε σχέση με την ατζέντα. Αν υπάρξει ξαφνικά μια κρίση, οικονομική ή άλλη, υπάρχει κίνδυνος να επισκιαστεί η άμυνα αλλά ελπίζω ότι θα υπάρξει αυτή η συζήτηση και το πρόγραμμα είναι ότι το, θα αρχίσει το Συμβούλιο με την συζήτηση της ασφάλειας και άμυνας. Θα είναι στην αρχή του προγράμματος. Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι η συζήτηση αυτή να μην είναι μια και έξω. Ο κύριος Ντονζόν είπε σωστά, δικαίως, ότι ίσως να μην υπάρξουν θεαματικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, αλλά αν κατορθώσουμε να κρατήσουμε την ασφάλεια και άμυνα στην ατζέντα των ηγετών μας, αυτό θα είναι ένα αποτέλεσμα ήδη που θα αξίζει. Ελπίζουμε να αρχίσει η διαδικασία, ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θα αναθέσει ορισμένες εργασίες στην ΕΠΑ το εκπρόσωπο, στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Εξωτερική, στην Υπηρεσία Εξωτερική εξωτερικής δράση για την ανάπτυξη δυνατοτήτων, διάφορα προγράμματα για τον οργανισμό, περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των αγορών άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε ε, να δώσει μια κατεύθυνση στο μέλλον. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Αυτό θα αποφασιστεί ούτω ώστε οι ηγέτες να μπορέσουν να αναθεωρήσουν ε, την κατάσταση και να εκτιμήσουν την πρόοδο που θα έχει ε, εκπληρωθεί. Στην έκθεση είπατε εκπρόσωπος περιλαμβάνει ιδέες για έναν χάρτη πορείας μακροπρόθεσμο για συνεργασία με στόχους και προθεσμίες. Θα πρέπει βεβαίως να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, αλλά αν ε, υπάρξει καλή συζήτηση και αν κατά κάποιο τρόπο υπάρξει ένας χάρτης πορείας και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορέσει να εγκρίνει ένα τέτοιο χάρτη πορείας ούτως ώστε η ασφάλεια και άμυνα να γίνει ένα θέμα που θα επανέρχεται συνεχώς στις συζητήσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Για να συνοψίσω, ε, τώρα είμαστε στην τελευταία ευθεία γραμμή πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση μία και έξω. Οι προτάσεις επιτάπητος μπορεί να μην είναι τόσο φιλόδοξες όπως ορισμένες προτάσεις που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι ε, πιο φιλόδοξο όργανο, αλλά ίσως δεν θα είναι επανάσταση, αλλά δεν θα είναι στασιμότητα. Δεν θα είναι μια στάσιμη κατάσταση. Θα υπάρξει πρόοδος και, ε, και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω πρόοδου για πολλά θέματα. Όταν δούμε ε, ποιες ήταν ε, οι αρχές των συζητήσεων στην αρχή του χρόνου, θα δούμε ότι διανύσαμε αρκετό δρόμο και ότι, υπάρχουν ε, σαφείς, ότι υπάρχει σαφής θετική δυναμική, όπως είπα και στην αρχή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δέσμευση, χρειαζόμαστε να τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν ότι τους ανήκει αυτή η πολιτική, να οικειοποιηθούν αυτή την πολιτική, Δελειώς δεν θα πάμε πολύ μακριά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι, σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ποπόφσκι. Αντίθετα ε, από όσα σας είχα πει θα ακούσουμε την κυρία Κλόντ Σαχνού ε, επικεφαλής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, εφόσον οι δύο αυτές παρουσιάσεις σχετίζονται με το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και νομίζω ότι αυτοί από εσά που ζήτησαν το λόγο θα ήθελαν να αντιδράσουν σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του Συμβουλίου. Καλύτερα να έχουμε μια συνολική, μια πλήρη ε, θεώρηση που θα, με την παρουσίαση που θα μας ε, παρουσιάσει σχετικά με τον οργανισμό. Κλοντ Φρανς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε δεχθεί μια αντιπροσωπεία στην υπηρεσία μας από ένα κράτος μέλος και δεν μπόρεσα να φύγω νωρίτερα. Αυτά που θα πω ίσως να έχουν ήδη υποθεί λοιπόν και θα τα επαναλάβω. Αυτό είναι προβληματικό. Από την άλλη αυτό θα δείξει ότι υπάρχουν και συγκλήσεις και ιδιαίτερα αυτόν τον τομέα στον οποίο ε, θα σταθούμε σήμερα οι συγκλήσεις είναι όλο και πιο έντονες πλησιάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το οποίο όλοι περιμένουμε ένα ισχυρό μήνυμα στα πλαίσια της στρατηγικής προβληματικής στην οποία βρισκόμαστε το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας είναι ζωτικό κατά προτεραιότητα σε ένα τόσο δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των δαπανών στον τομέα της άμυνας και η μεγιστοποίηση της προσπάθειας στον τομέα της άμυνας είναι κάτι που περνάει από τη συνεργασία, είναι κάτι το οποίο περνάει από την χρήση των μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από συνέργειες με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μία μόνιμη εμπλοκή θα έλεγα και των αρχηγών κρατών και των αρχηγών κυβερνήσεων να επανέρχονται στο θέμα και να επανέρχονται στις προτεραιότητες τις οποίες έχουν θέσει και στους προσανατολισμούς τους οποίους έχουν ορίσει για τις διαφορετικές δομές της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η ευθύνη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι φυσικά η ασφάλεια των πολιτών και η χρήση των ενόπλων δυνάμεων. Είναι το θέμα δηλαδή της κεντρικής ευθύνης την οποία έχουν τα κράτη-μέλη. Τα θέματα αυτά προσπαθούμε λοιπόν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να το θέσουμε ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο ΝΑΤΟ απαιτείται συγκλήσεις γύρω από αυτό αλλά θέτοντας το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θα έλεγα ο καλύτερος χώρος συνδυασμού και των οικονομικών υποχρεώσεων, κατά συνέπεια και των δημοσιονομικών υποχρεώσεων και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν την προτεραιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει τα θέματα της άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν να διαιτητεύσει κανείς υπέρ των δαπανών για την άμυνα. Εδώ είστε αρμοδιότεροι εμού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδέα σύμφωνα με την οποία η στρατιωτική δράση σε πολλές περιπτώσεις παραμένει μία επιλογή. Μπορεί να βασιστεί κανείς όσο μπορεί περισσότερο στην πρόληψη. Μπορεί να καλλιεργήσει τις συνέργειες οι οποίες δημιουργούνται σε επίπεδο κράτους δικαίου κατάρτισης, εκπαίδευσης, παιδείας. Αυτά όλα είναι κεφαλαιώδη, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει η άλλη δυνατότητα από τη χρήση βίας ή από την έστω, δυνητική χρήση βίας σε επίπεδο απειλής. Λοιπόν, η χρήση βίας παραμένει σαν μια επιλογή ή η απειλή χρήση βίας. Καμία πολιτική πρόληψης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ύπαρξη της στρατιωτικής δύναμης και της δυνητικής χρήσης της. Στο εσωτερικό αυτής της ικανότητας της στρατιωτικής θα πρέπει να είμαστε επίσης ε, ε, απαιτητικοί σε επίπεδο αρκτικό, σε επίπεδο θα έλεγε κανείς έναρξης της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείχνουν ότι είναι σε θέση να αναλάβουν μία αποστολή ε, εφόσον έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Βέβαια πρέπει να επιδείξουν την επιθυμία να το κάνουν και αυτό είναι μια πρώτη προϋπόθεση. Πρέπει οι Ευρωπαίοι λοιπόν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ικανοί σε περιπτώσεις κρίσης να θέσουν τις δυνάμεις τους, να τις καταστήσουν διαθέσιμες έτσι ώστε να μπορέσουν οι περιφερειακές οργανώσεις ή κυρίως τα Ηνωμένα Έθνη να χρησιμοποιήσουν τις πολιτικές και στρατηγικές δυνατότητες τις οποίες τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να προηγηθεί. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν λοιπόν, πρέπει να ληφθούν άμεσα στον τομέα συγκεκριμένων δράσεων έτσι ώστε να υπάρξει σωστή χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων. Όλοι συνειδητοποιούμε βέβαια ότι το μήνυμα προέρχεται από τους βασικούς μας εταίρους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν υπάρχει α, δυσ, ε, δυσαρμονία ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Περιμένουν οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως security provider, παροχέας ασφαλείας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και αυτό το οποίο συμπεριέλαβε η Κάφη Άστον στην έκθεσή της ως ύπατη εκπρόσωπος αλλά και ως υπεύθυνη της δικής μας υπηρεσίας είναι να προσπαθήσει να συγκεκριμενοποιήσει το μήνυμα αυτό με συγκεκριμένα προγράμματα ακριβώς έτσι ώστε να καλυφθούν οι ικανότητες που ελείπουν σήμερα και κάποια πρακτικά κίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν σε καλύτερες μορφές συνεργασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων για τις ικανότητες της στρατιωτικές. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο Ματιό. Ξέρετε ότι ανεφοδιασμός εν πτήση είναι ένα βασικό πρόβλημα και κενό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, κάλυψαν το 80% των ε, αναγκών που είχαμε σε επίπεδο ε, τροφοδοσία σε καύσιμα εν πτήση. Σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας προσπαθήσαμε να εργαστούμε και σε επίπεδο βραχυπρόθεσμο και σε επίπεδο μεσοπρόθεσμο και σε επίπεδο μακροπρόθεσμο. Σε επίπεδο βραχυπρόθεσμο προσπαθήσαμε να μεγιστοποιήσουμε την δυνατότητα της Ιταλίας σαν παράδειγμα. Έχει ε, ανεφοδιαστικά αεροσκάφη τύπου Boeing 767 και να συνδυάσουμε τις δυνατότητες των, Ιταλικών αεροσκαφών ε, και των ε, καταρτικών άλλων χωρών όπως η Σουηδία και η Γαλλία και να προσπαθήσουμε να πιστοποιήσουμε την δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά αεροσκάφη πολεμικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, σύντομα το α400 μ της ΕΡΒΑΣ... και σαν μεταγωγικό και σαν ανεφοδιαστικό καυσίμων εν πτήση. Απαιτείται να υπάρξει ένας στόλος πολλαπλών ρόλων αεροσκαφών ανεφοδιασμού και ανεφοδιαστικά και μεταφορικά και ε, εκενώσεις σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, τα λεγόμενα δηλαδή αεροσκάφη MRTT, πολλαπλών ρόλων αεροσκάφη και επίσης δυνατότητα συζήτησης από εδώ και πέρα για από κοινού αγορά τέτοιου, είδου είδους αεροσκαφών με προγράμματα τα οποία βλέπουν ότι κάποιες χώρες θα αποκτήσουν νέα ανεφοδιαστικά αεροσκάφη όπως το Voyager στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν στο μέλλον για την απόκτηση τέτοιου είδους αεροσκαφών και βραχυπρόθεσμα να δράσουμε και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα πραγματικό στόλο ανεφοδιαστικών αεροσκαφών. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, καθοριστικό, θα το πω αγγλικά. Είναι τα λεγόμενα remotely pilot ε, aircraft, δηλαδή ε, μακρόθεν καθοδηγούμενα αεροσκάφη, τα λεγόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones με ε, μια σύντομη έκφραση. Αυτή η μελλοντική γενεά των drones θα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές χρήσεις. Ε, τα drones θα χρησιμοποιούνται και για μη στρατιωτικούς λόγους αλλά και για στρατιωτικούς λόγους. Έχουν διεισδυτική ικανότητα στο σύνολο του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου και θα πρέπει εδώ να ρυθμίσουμε και τα θέματα τα ρυθμιστικά που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξαρτώνται από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις τεχνολογικές πλευρές, τα θέματα ασφαλείας για την κυκλοφορία, την ασφαλή των μη επανδρομένων αεροσκαφών και φυσικά το στρατιωτικό κομμάτι, την προετοιμασία, την προπαρασκευή της επομένης γενεάς μη επανδρομένων αεροσκαφών, έτσι ώστε να αυξήσουμε την δυνατότητά τους και να χρησιμοποιήσουμε εν τω μεταξύ τις παρούσες ικανότητες τις οποίες αποκτούν σταδιακά ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αρκετά θέματα λοιπόν στα οποία πρέπει να προχωρήσουμε, το ρυθμιστικό διακανονιστικό, το τεχνολογικό και οι μελλοντικέ εξελίξεις συνεργαζόμενοι παράλληλα με βάση τους υπάρχοντες εξοπλισμούς. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι σε επίπεδο διαστημικής πολιτικής να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο θέμα φυσικά των δορυφόρων τηλεπικοινωνιών και την προετοιμασία των επομένης γενεάς ε, ε, διασφαλισμένων σε επίπεδο αν θέλετε εμπιστευτικότητας και χρήσης ε, τέτοιου είδους σκαφών στο διάστημα. Υπάρχει επίσης και ο τομέας της κυβερνοασφάλειας εδώ θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο κυβερνητικής άμυνας ή κυβερνοάμυνας να το πω καλύτερα. Κοινή έρευνα και ε, προσπάθεια για νέες τεχνολογίες με προστασία των ε, αποστολών μας, των εγκαταστάσεών μας, των βάσεών μας, των στρατηγίων μας κτλ. Και αυτό το κάνουμε βέβαια σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και με δορυφορικούς τρόπους. Συναντήθηκα με εκπροσώπους πρόσφατα από την Εσθονία που είναι μια από τις ηγέτιδες χώρες, έχουν πάρα πολλές και καλές ιδέες στον τομέα της κυβερνοπροστασίας για τα επόμενα χρόνια. Έχουν, λοιπόν, περιμένουμε αποφάσεις στη Διαχειριστική Επιτροπή της Υπηρεσίας και από πλευράς ε, των ε, Υπουργών Άμυνας έτσι ώστε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επί τη βάση των προπαρασκευασμένων αποφάσεων να μπορέσουν να προχωρήσουν ε, στην εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. Πέρα από τα ειδικά προγράμματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας αυτό το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα συνεργασία μας. Στον προηγούμενο χρόνο υπεγράφει ένας κώδικα συμπεριφοράς για την προσφυγή στην συνεργασία. Οι κυβερνήσεις στο δικό τους επίπεδο μπορούν να εφαρμόσουν τον κώδικα αυτό σε εθνικό επίπεδο. Όταν λέμε σε αυτόν τον κώδικα, σαν παράδειγμα, ότι τα προγράμματα συνεργασίας είναι η προτιμόμενη επιλογή για την διασφάλιση μιας στρατιωτικής ικανότητας και είναι και προγράμματα τα οποία θα πρέπει να προστατεύσουμε κατά προτεραιότητα από τις δημοσιονομικές μειώσεις. Πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης να γίνει πραγματικότητα. Θα πρέπει να εργαστούμε επίσης και στα διαφορετικά επίπεδα τα οποία συντελούν στην συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή φορολογικά και ε, χρηματοοικονομικά θέματα. Υπάρχει επίσης και μια σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της ανακοίνωσης την οποία δημοσίευσε πρόσφατα. Πρέπει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να δώσουν προσανατολισμούς στα θεσμικά όργανα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις υπόλοιπες δομές όπως η Υπηρεσία Άμυνας, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τις ισχύουσες συνέργειες σήμερα. Οι συνέργειες αυτές σε ορισμένους τομείς μπορεί να είναι βασικές στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, σαν παράδειγμα. Αυτό υπογραμμίστηκε και σε πολλές δικές σας εκθέσεις, και σε επίπεδο βέβαια κοινοβουλίου, αλλά και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Εμείς φοβάμαι ότι διακινδυνεύουμε οριακά στην παρούσα φάση την υπεροχή, την τεχνολογική η οποία μας χαρακτήριζε μέχρι τώρα και η οποία ήταν ζωτική για την ευημερία μας. Θα πρέπει ότι είναι διοικού χαρακτήρα δομές να αντιστηρίξουμε με συνέργειες ανάμεσα στα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και άλλες πηγές πιθανώς χρηματοδότησης, τις οποίες το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να εντοπίσουν. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε κάποιες τέτοιες πηγές διπλής χρηματοδότησης, διτής αν θέλετε χρηματοδότησης, χωρίς όμως να θέσουμε σε αμφισβήτηση την υπεροχή μας στον τομέα της τεχνολογίας. Όταν μειώνουμε τα δημοσιονομικά, το πρώτο το οποίο μειώνουν τα κράτη-μέλη είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, γιατί εκεί μπορούν άμεσα να μειώσουν το κόστος χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερα υψηλό πολιτικό κόστος μετά από τις αποφάσεις τους. Ένας άλλος τομέας είναι αυτός ο οποίος έχει σχέση με την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπως λένε οι ίδιοι εκπρόσωποι της περνούν από προγράμματα, από χρήματα, από χρονοδιαγράμματα. Περνούν επίσης και από την στήριξη ορισμένων οριζοντίων μέσων. Ό,τι μπορεί να υπάρξει ανάμεσα την δική μας υπηρεσία και τις ε, μικρομεσαίες και μεσαίες ενδιάμεσες επιχειρήσεις είναι τομέα στον οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Για να είμαι σύντομη, ε, στον τομέα των συνεργειών, στα πλαίσια της διευρυμένης ευρωπαϊκής οικογένειας μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία συνεργαζόμαστε με την Διαστημική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία με το ΝΑΤΟ φυσικά και η συμπληρωματικότητα εδώ με το ΚΑΡ και το λέει αυτό και στην έκθεσή του ο κύριος Γκάλερ υπάρχει η δυνατότητα ε, να υπάρξει σύγκληση μέσω του διαχειριστή προγραμμάτων που είναι το ΚΑΡ εργαστήκαμε και σε προγράμματα τα οποία επιτρέπουν να προστατεύσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή των κοινοβουλίων και να υπάρχει φυσικά κοινή χρήση των δυνατοτήτων. Σαν παράδειγμα κοινό στρατηγείο για τις αεροπορικές μεταφορές, ε, τις εννοούμε σε στρατιωτικό επίπεδο. Ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαβηνθεί και σε άλλους τομείς. Ίσως έχω μακρηγορήσει, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Προσπαθήσαμε λοιπόν στην παρούσα φάση να τροφοδοτήσουμε τις συζητήσεις του Συμβουλίου για τα θέματα της άμυνας. Πρέπει να επιστρέψουμε και να τα συζητήσουμε αναλυτικά, να δείξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, γιατί η άμυνα είναι προτεραιότητα και πρέπει η προσπάθεια γύρω από την άμυνα να είναι αποτελεσματική. Αυτό θα αποδειχθεί από συγκεκριμένα κίνητρα, από συγκεκριμένα προγράμματα. Κάποια από τα προγράμματα αυτά δεν έχουν πάρει την τελική τους φάση σήμερα ε, και όπως είπε ο Ματιό θα μπορέσουν να ε, οριστούν καλύτερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του επερχόμενο. Υπάρχουν προσδοκίες και πρέπει να υπάρξουν και απαντήσεις που να καλύψουν τις προσδοκίες και του κοινού και των εμπλεκομένων, δηλαδή επιχειρήσεων, στρατιωτικών ηγεσιών κτλ. Σας ευχαριστώ Κλοντ Φρανς, ιδιαίτερα πλήρης η παρέμβασή σας. Θα υπάρξουν αρκετές αντιδράσεις, έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Θα ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων πρώτο. Μπόγκταν Κλίσ από την Πολωνική Γερουσία, τέος Υπουργός Άμυνας. Κύριος Κλίσ. Ε, σας ευχαριστώ. Στην αρχή, εκ θα ήθελα να τονίσω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης του τελικού αποτελέσματος ε, του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η τρίτη φορά που συναντόμαστε εδώ από όσο θυμάμαι και που συζητάμε τα θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της κοινή πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η τελική έκθεση που προσφάτως δημοσιεύθηκε θεωρώ ότι περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές διατάξεις. Ένα ωστόσο είναι σημαντικό. Μία άποψη η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη συμφωνημένη συμφωνημένο όραμα για το μέλλον της ΚΕΠΑ. Αυτά αναφέρει δηλαδή Άστον στην έκθεση. Το καταλαβαίνω αυτό πολύ καλά. Καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια πρόκληση για ε, το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά και για όλες τις μελλοντικέ μας δραστηριότητε και μετά από το Συμβούλιο. Να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις τώρα, σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, πολιτικής ασφάλειας Καταρχάς ε, σε ό,τι αφορά την ενοποίηση των δύο πολιτικών αυτών. Στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει ε, πολύ συνεκτική ε, πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο της Ένωσης. Να μην βασίζεται στα συμφέροντα κάποιων σημαντικών κρατών μελών, αλλά στα συμφέροντα της ασφάλειας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο. Κατά δεύτερον, αυτή η ενοποίηση των δύο αυτών μέσων σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο ανοιχτή προσέγγιση. Αυτό τι σημαίνει ότι πολιτικά, ε, διπλωματικά, οικονομικά θα πρέπει όλα τα μέσα να δημιουργούν μια ευρύτερη πολιτική προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φυσικά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία έτη στους τομείς αυτούς ε, και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο κέρας της Αφρικής. Πολλά ωστόσο παραμένουν ακόμα εκρεμή πρώτη παρατήρηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δυναμικού. Θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω ε, εξέλιξη της δραστηριότητα αυτής της ε, ενοποίησης αυτής. Θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω ε, αξιοποίηση των εφιστάμενων δομών, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, το σχέδιο ανάπτυξης δυναμικού, η τεχνολογική και βιομηχανική βάση εκ παραλίλου, η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, ξεχωριστό κεφάλαιο. Αυτή η εναρμόνιση, είμαι σχετικά βεβαίως, θα πρέπει να ενδυναμωθεί σε διάφορα επίπεδα STM e και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας του προγράμματος Pooling and Sharing και του προγράμματος Ευθύους ε, Άμυνας αλλά ιδιαίτερο μεταξύ της υπηρεσία και του ACT e σε ό,τι αφορά το δυναμικό. Τώρα, τέταρτη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τις ε, επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο έντονα στον τομέα αυτό. Καταρχάς, επειδή έχουμε συγκεκριμένα επιτεύγματα που είναι σαφή. Κατά δεύτερον, επειδή υπάρχει κρίση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το μαλλί. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την διάθρωση των μέσων αυτών και να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνιμου, μόνιμες τέτοιες ικανότητες. Κατά δεύτερο, να προωθήσουμε πολυεθνικές λύσεις σε ό,τι αφορά κρίσιμες δυνατότητες. Αναφέρθηκα ήδη στο pooling and sharing. Και κατά τρίτο, να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στα battle groups, groups ομάδες αυτές μάχης να εξετάσουμε περαιτέρω λοιπόν το θέμα αυτό πέρα από την ε, έκθεση, αυτό που προτείνει η έκθεση της είπα της εκπροσώπου. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλά έχουμε πετύχει, μεγάλα επιτεύγματα έχουμε πετύχει, αλλά πολλά παραμένουν ακόμα μπροστά μας, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αξιοποιήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση το πλήρες δυναμικό μας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και για φλέπω το CFTP θα πρέπει να μας δώσει πιο πολλές δυνατότητες για τις οργάνωση, για τον συντονισμό, το στρατιωτικό και στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Αρχηγείο θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα και μόνο προς τα επιχειρησιακό στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω μία μέρα να ζήσουμε και να δούμε την δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Η CFTP δεν χρειάζεται νομίζω καινούργιες δομές, αλλά πολιτική βούληση και ένα νέο κίνητρο, ένα νέο σπρόξιμο αν θέλετε, όπως πριν από εννέα χρόνια που δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ σημαντική ευρωπαϊκή στρατηγική και την πρώτη σημαντική τέτοια ευρωπαϊκή επιχείρηση της Αλθέα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια, ένα μακρύ όραμα για την ανάπτυξη του CSDP. Ευχαριστώ πολύ Μπογκδάν. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Έλιο Βίτε από το, την Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων. Καλημέρα Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, οργάνωση αυτής της συνάντησης της διακοινοβουλευτικής. Είναι μια περαιτέρω ευκαιρία για μας για τη σωστή αξιοποίηση των ρόλων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταστήσουμε πιο διαφανείς τις αποφάσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας. Όπως ε, είπαμε για τη συνάντηση στο Βίλνιον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια απλή μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις στα πλαίσια του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, είναι συνδυασμός εθνικών κυριαρχιών και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν πιο θαραλέες αποφάσεις στο πλαίσιο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή δράση χωρίς την πολιτική ένωση. Αυτή η πολιτική ένωση λοιπόν είναι το επόμενο ευαίσθητο βήμα στο οποίο θα πρέπει να περάσουμε και προς το οποίο οδεύουμε. Μια ενωμένη Ευρώπη σε πολιτικό επίπεδο θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σε υπηρετικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια του Συμβουλίου του μηνός Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσουμε τις δυνατότητες ε, τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Άμυνα, να αναπτύξουμε τις δυνατότητες αυτές ακόμα περισσότερο και στον πολιτικό και στον στρατιωτικό τομέα. Να προωθήσουμε τις βιομηχανικές συνέργειες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυξάνοντας τον βαθμό συλλογικής ασφαλείας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκτώντας μεγαλύτερη εξουσία, σε εισαγωγικά αν θέλετε, σε διεθνές επίπεδο. Να προσπαθήσουμε να έχουμε την δυνατότητα άμεσης απόκρισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν χρειάζεται, να επιμερίσουμε σωστά τους υπάρχοντες πόρους, να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας έτη περαιτέρω και να προωθήσουμε τη βιομηχανική συνεργασία έτσι ώστε να μην συνεχιστεί η πορεία προς την παρακμή. Αυτά τα θέματα δεν είναι, θα έλεγε κανείς, καινοτόμα σαν σε επίπεδο παρατήρησης, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Στην προηγούμενη συνάντηση του Βίλνιους είπαμε ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να κινητοποιήσουν τη συζήτηση στον τομέα της ασφάλειας, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας από πλευρά των πολιτών και να υπάρξει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών πιστεύω για να εργαστούμε σε επίπεδο μεθοδολογικό πλέον και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και εδώ θα κάνω κάποιες προτάσεις. Σε επίπεδο μεθοδολογίας τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια θα πρέπει να προχωρήσουν σε πράξεις κατευθυντήριες προς την πλευρά των κυβερνήσεών τους έτσι ώστε να προσανατολίσουν σωστά τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να χαρακτούν ορισμένοι κοινοί προσανατολισμοί, κοινοί παρανομαστές, αναπόσπαστο τμήμα της κάθε χώρας και σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας προς τους πολίτες, έτσι ώστε να αναγνωριστεί και η μη στρατιωτική διάσταση της ΚΕΠΑ ιδιαίτερα σε σχέση με τις δομές οι οποίες έχουν σχέση με την πρόληψη των κρίσεων για τη δική μου χώρα, την Ιταλία. Και τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα εδώ και μήνες εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια ορισμένων ανιχνευτικών ερευνών, οι οποίες έχουν σαν στόχο να εμπλουτίσουν τις συζητήσεις του Συμβουλίου τον μήνα Δεκέμβριο. Αυτές τις ημέρες προστίθεται και η διαδικασία μεταρρύθμισης των, πολι... πολεμικών στρατιωτικών μάλλον σχηματισμών στην χώρα μου και η γνωμοδότηση της Ιταλικής Βουλής η οποία είναι δεσμευτική θα εκδοθεί τον μήνα Νοέμβριο. Θα επιβεβαιωθεί επίσης και η απόφαση ε, της κυβέρνησης για την συνέχιση της χρηματοδότησης των ειρηνευτικών αποστολών. Οι συζητήσεις που θα γίνουν γύρω από αυτό είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επιστήσουν την προσοχή της κοινή γνώμης της Ευρωπαϊκής στα θέματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Η Ιταλία έχει και μια συγκεκριμένη ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων οι οποίες θα ληφθούν. Ε, το εξάμεινο προεδρίας της θα ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εκλογές και θα είναι μια νέα φάση ανανέωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ της Και γι' αυτό ακριβώς συμμετέχουμε στην σημερινή συνάντηση με πάρα πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται μετά το Βίλνιος... να συνομιλήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θεωρώ ότι αυτό γίνεται και εγκαίρως πριν τη διεξαγωγή του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ήσασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, κυρία Νου, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα, τα συγκεκριμένα project τα οποία αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι από αυτό καθίσταται σαφές ότι πολλά υπάρχουν, πολλά υπάρχουν τα οποία χρειαζόμαστε να τα κάνουμε από κοινού και τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Ούτε χρειάζεται. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο Συμβούλιο να ασχοληθούμε, να ενσκύψουμε πάνω σε τέτοια θέματα στους τομείς εκείνους όπου συμφωνούμε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε πλέον από την ε, παραδοσιακή, αν θέλετε, ε, και αποκλειστικά εθνική θεώρηση των θεμάτων αυτών. Θεωρώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει πραγματικά να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις τους προκειμένου να αναπτυχθούν νέες δομές και νέες νοτροπίες στα εθνικά Υπουργεία Άμυνας, στα, στις εθνικές υπηρεσίες εξοπλισμών. Αυτό λοιπόν, ε, σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να σκεφτούμε ευρωπαϊκά, γιατί ε, παραδοσιακά επικρατεί ένας εθνικός τρόπος σκέψης, αλλά αυτό πλέον δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Μιλάμε για κάποιους τομείς, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν υπερβολικές, υπερβολικά υψηλές ικανότητες και δυνατότητες και σε άλλους τομείς ε, υπάρχουν μεγάλα κενά. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν παραγωγή, άρα γίνεται αγορά. Γίνονται αγορές ε, σε κάποιες τυχαίες χώρες, ενώ άλλες χώρες που παράγουν τελικά δεν έχουν αρκετή ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι στο Συμβούλιο θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα συνεργασίας βιομηχανικής, αλλά και τους κανόνες που έχουμε στον τομέα της τυποποίησης, της πιστοποίησης, να δοθεί μια όθηση προκειμένου από κοινού να κάνουμε πιο πολλά. Να ερωτήσω προς τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και κυρίως όχι στα κοινοβούλια, αλλά στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις υπηρεσίες ε, εξοπλισμού. Εσείς είσαστε έτοιμοι να προασπίσετε αυτή την καινούργια ανατροπία, προκειμένου να αρθούμε στο ύψος των ε, περιστάσεων. Ελπίζω αυτό το Συμβούλιο να αποτελέσει μια πρώτη τέτοια ευκαιρία και να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία να καταλήξουμε σε κάποια κοινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στο συνάδελφο από την Πορτογολία, Μιράντα Κάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ, πρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΕΤ, για την πρόσκλησή του και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Βάντρομπει και τον κύριο Μάρτιν Σούλτς για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τα θέματα αυτά. Κατά πρώτο λόγο νομίζω ότι όσον αφορά στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να υπάρξει ευθύς εξ αρχής ένα κονσένσους, μια γενική συνένεση. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια στρατηγική ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά αυτή ε, χρονολογείται από το 2003 αναθεωρήθηκε το 2008, αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει και πάλι να αναθεωρηθεί εκ για να ληφθούν υπόψη ε, διάφορα στοιχεία, η μετεξέλιξη στο ΝΑΤΟ κλπ. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα κονσένσου σχετικά με αυτήν την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Δεύτερον, η συνεργασία. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας πάρα πολύ συχνά χαρακτηρίζεται από κατατεμαχισμό των θέσεων σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν πρωτόκολλα διμερεί συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημειακές κατά περίπτωση πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σχετικά με την άμυνα και γνωρίζουμε ότι σε ένα πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ορισμένα προβλήματα ε, και σκέφτομαι τη Λιβύη, το Μαλί ε, και τη Συρία. Πρόσφατα μιλήσαμε επίσης για την ορατότητα, το πόσο γνωστή είναι αυτή η πολιτική. Πήγα σε ένα στρατόπεδο προσφύγων, σύρων προσφύγων στην Τουρκία και πάρα πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες με ρώτησαν πού είναι η Ευρώπη, πού βρίσκεται η Ευρώπη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβη σχετικά με τη Συρία και την πολιτική σε σχέση με τη Συρία. Έχουν ληφθεί σημειακές αποφάσεις οι οποίες είναι η απόδειξη μιας πραγματικού κατατεμαχισμού των θέσεων. Δεν υπήρξε ε, θέση και πρόπτικη κοινή σε σχέση με τη Συρία και σύνεπώς όταν μιλούμε για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχει κάποια, θα υπάρξει κάποια ευελιξία στις θέσεις. Είναι ουσιαστικό αυτό. Είναι ουσιαστικό να αναγνωρίσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών μας, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αναγκαιότητα να προωθήσουμε την συνεργασία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι αντίθετα με τα όσα πιστεύουμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι στα θέματα αυτά αρκεί να σκεφτούμε το τι συμβαίνει στη Λαμπεντούζα με την άφηξη προσφύγων από τη Βόρεια Αφρική. Και η στρατηγική δεν είναι σαφής εκεί ως προς τους πρόσφυγες και ως προς την ασφάλεια συνεπώς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ευελιξία, ε, συντονισμός και κάποια ευελιξία στο συντονισμό, ούτω ώστε ε, για να έχει μια καλή βάση αυτή η μελλοντική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στο θέμα ε, της, της βιομηχανίας, της τη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτών των βιομηχανιών, αλλά θα πρέπει πολλοί τομείς να συνδεθούν με αυτήν την ανάπτυξη. Ο τομέας, οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν πολλές θέσεις εργασίας στις χώρες μας και εδώ υπάρχουν δύο Ευρώπες, διότι δεν βλέπω καμία ορατότητα, να υπάρξει καμία ορατότητα σε επίπεδο βιομηχανικό σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα αλλά υπάρχει μια ορατότητα της Ευρώπης, του Eurogroup όσον αφορά στα θέματα τα οικονομικά και τα χρηματοπιστωτικά. Το Eurogroup που μας επιβάλλει πολιτικές λιτότητας. Εκεί είναι πολύ ορατή η Ευρώπη. Σε άλλους τομείς θα πρέπει να είναι εξίσου ορατή η Ευρώπη. Όσον αφορά στην ασφάλεια και στην άμυνα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίως ε, τις δημοσιονομικές απόψεις, αλλά δεν θα πρέπει να αρνηθούμε την ε, σημασία, να απορρίψουμε τη σημασία της ασφάλειας και της άμυνας και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δύο Ευρώπες. Υπάρχουν χώρες που έχουν την δική τους αμυντική βιομηχανία, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στον οικονομικό τομέα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον οικονομικό τομέα. Αν δεν υπάρξει ισορροπία, θα βρεθούμε απομονωμένοι και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα που έχουμε ήδη αυτή της δημοσιονομικής λιτότητας που έχει επίσης συνέπειες για τον προναμιντικό προϋπολογισμό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα δημιουργήσουμε ένα νησί για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυκτό. Είπα ότι η εκπρόσωπος κυρία που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να θεσπίσει μια πολιτική για τη συμπερίληψη όλων αυτών των τομέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να προβλεφθούν επίσης στο μέλλον προϋπολογισμοί κατάλληλοι για την ασφάλεια και την άμυνα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς θα πρέπει να εφαρμόσω τον χρόνο ομιλία στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελειώς δεν θα έχουμε απάντηση από τους παρουσιαστές και που θα, θα είναι κρίμα και το σύνολο των συμμετοχόντων δεν θα μπορέσουν να λάβουν τον λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι, τρία λεπτά maximum για τον κάθε παρεμβαίνοντα. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντελπικά της Γαλλικής Γερουσίας. Τρία λεπτά, αγαπητοί συνάδελφοι, σε τρία λεπτά θα κάνω πέντε παρατηρήσεις. Πρώτον, η απόφαση συμπερίληψης της άμυνας στην ημερήσια διάταξη του το Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που θα, ε, ε, που θα συνεδριάσει σύντομα είναι πάρα πολύ καλό. Σας συγχαίρω γι' αυτό. Ε, περιμέναμε πέντε χρόνια για να ξαναγίνει λόγος για το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο βλέπουμε είμαστε αδύναμοι μπρος την πτώση των αμυντικών δαπανών λόγω οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών της συνεπειών. Τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την κρίση, να την θεωρήσουν ευκαιρία για να ενωθούν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Τρίτον, υπάρχει σε αυτήν την ε, ε, σε αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα θέματα άμυνας ενώ η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται υπάρχει σε αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος ένα ε, θέμα που οδηγεί να θυσιάζονται οι ένοπλες δυνάμεις για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχει έλλειψη απειλής για την κοινή γνώμη και επίσης επικάλυψη του ΝΑΤΟ. Αλλά ο λόγος ο βασικός που εμποδίζει κάθε πρόοδο σήμερα προς μια αυθεντική ευρωπαϊκή άμενη είναι το θέμα της κυριαρχίας. Έχει το όνομα κυριαρχία. Οι ευρωπαϊκές ε, κυβερνήσεις προσπαθούν, ε, προτιμούν να εξαλειφθεί η αμυνά τους παρά να παραχωρήσουν κυριαρχία. Τέταρτον, αυτό δεν ωφελεί σε τίποτα να κάνουμε διαμαρτυρίες υπέρ μιας λευκής βίβλου ή μιας βάσης βιομηχανικής και τεχνολογικής για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, ενώ θα υπάρχει αυτό το θέμα της κυριαρχίας. Ο λόγος είναι απλός. Αυτό που λείπει είναι ένα όργανο, ένα όργανο διαιτησίας που να μπορεί να αποφανθεί, να δώσει μια απάντηση σε διάφορες διαφωνίες σε αποκλίνουσες απόψεις. Αν θέλουμε πράγματι να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Άμυνα, θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε το θέμα της κυριαρχίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Γαλλική Γερουσία ε, εκπώνησε μια σύντομη έκθεση τον Ιούλιο με τίτλο «Για να τελειώσουμε με την Ευρώπη της άμυνας προς μια αυθεντική ευρωπαϊκή άμυνα». Και έχω εδώ μερικά αντίγραφα αυτή της έκθεση στη διάθεσή σας, ακόμα και στα αγγλικά. Βλέπετε λοιπόν ότι κάνουμε το παν για να εξηγηθούμε καλά. Τι θέλουμε, ποια είναι η σύστασή μας. Η σύστασή μας είναι ότι θα πρέπει να συγκροτήσουμε ένα Eurogroup άμυνας. Επαναλαμβάνω, ένα Eurogroup άμυνας ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν και μπορούν μέσα στην οποία ομάδα δεν θα ισχύει πλέον ο κανόνας της ομοφωνίας. Έτσι η Ευρώπη προχώρησε κάθε φορά για το νόμισμα, για το ευρώ, για τα σύνορα, Schengen και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Ίσως αυτό να φαίνεται όνειρο σε μερικούς, αλλά όπως έλεγε ο Σέπτσοξ, είναι αυτοί που είναι αρκετά τρελοί για να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, που θα τον αλλάξουν πράγματι. Και εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας είμαι λίγο επίοικης, ίσως θα, θα θεωρηθεί κακή η προαίρεση, διότι μιλήσατε 3 λεπτά 50 αντί για τα 3 λεπτά που είχατε στη διάθεσή σας. δεν υπάρχει εδώ μετρητής, αλλά νομίζω ότι αυτά που είχατε να πείτε νομίζω ότι άξιζαν τον λόγο. Νομίζω ότι η έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας αξίζει να διαβαστεί χωρίς ε, κανείς να εξαπατηθεί από τον τίτλο που δεν αναφέρεται ακριβώς στο περιεχόμενο. Δίνω στην ε, Μαρία Ελένη Κοπά που είναι η συγγήτριά μας Ευρωβουλευτής φέτος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας που θα παρουσιάσει την επόμενη Ολομέλεια την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που θα παρουσιαστεί πριν από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντική αυτή είναι η συζήτηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί εκεί, στα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, λαμβάνονται οι πραγματικές αποφάσεις ε, και θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ε, πολιτική ασφάλεια. Στο Νότο λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολε οι προσδοκίες και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολη η συζήτηση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνάει πολύ δύσκολες εποχές η Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες περικοπές, ιδιαίτερα στο θέμα της άμυνας. Άρα χρειαζόμαστε μια μεγάλη δέσμευση για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και Άμυνα είναι υψηλό το επίπεδο των προσδοκιών μας και των φιλοδοξιών μας, παρά το γεγονό ότι συχνά τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Με πολύ επικοδομητικό τρόπο έχουμε εργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε συνεργαστεί και με το Συμβούλιο. Έχουμε λάβει και πολύ αισιόδοξα μηνύματα από την Υπηρεσία Εξαιρετική Δράση, παρά το γεγονό ότι δεν είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξία τα μηνύματα αυτά. Άρα, θα πρέπει να συζητήσουμε για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι όντω τέτοιο πάροχο ασφάλεια ή θα εξακολουθήσει να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μεγάλη ώρα με κανένα άλλο παραπάνω ρόλο σε επίπεδο άμυνας Νομίζω ότι για όλους εξημών που είμαστε δεσμευμένοι για την κοινή πολιτική αυτή, το κλειδί είναι η συνεργασία, η ανάπτυξη α, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, θεωρώ. Κάποια σημεία να αναφέρω. Καταρχάς χρειαζόμαστε μια στρατηγική επικοινωνία. Οδεύουμε προς το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και ακόμα και σε συγκεκριμένα φόρα εδώ πέρα στο κοινοβούλιο, στις, στις επιτροπές, στα εθνικά κοινοβούλια όπου συζητάμε θέματα αμήνης δεν υπάρχει η ορατότητα που χρειάζεται για την ευρωπαϊκή αυτή συζήτηση που σχετίζεται με την ασφάλεια του πολίτη στη τελική ανάλυση. Θα πρέπει λοιπόν να τεθεί αυτό το θέμα στην ατζέντα των ευρωεκλογών. Κατά δεύτερον, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε παντού παρόντες. Πρέπει να επιλέξουμε τους στόχους μας, αλλά Τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε, να κάνουμε στρατηγικές επιλογές που δεν είναι πάντα, αν θέλετε, προφανείς και εύκολες. Τρίτον, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε που αναφέρεται στην έκθεση της ΕΠΑ της ε, εκπροσώπου, το θέμα της θαλάσσιας ε, ασφάλειας και της ασφάλειας των συνόρων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα και στην στιγμή που μιλάμε ε, γίνονται πολλά σημαντικά βήματα και Πραγματικά θα πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό μετά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου κατά τέταρτον, να αξιοποιηθεί στο έπακρον το δυναμικό που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο δεν γίνεται. Όσοι θέλουν να προχωρήσουν προς τα εμπρός να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και οι υπόλοιποι δεν θα πρέπει να τους παρεμποδίζουν, να τους παρακολύουν. Να εφαρμοστεί λοιπόν σωστά η συνθήκη, να εφαρμοστεί τα θέματα περί ταμείου, startup, αυτά που αναφέρονται για όλα τα θέματα αυτά. Κατά πέμπτον, οι σχηματισμοί αυτοί μάχη, τα battle groups, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν λύσεις που θα καταστήσουν αυτό το μέσο ε, ε, λειτουργικό και πιο ευέλικτο. Πώς θα δημιουργηθούν τέτοιες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Θα πρέπει να το συζητήσουμε όμως και μάλιστα ανοιχτά. Τέλος, το ΝΑΤΟ ασφαλώς. 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη και του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει λοιπόν οποιαδήποτε, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Ας συνεργαστούμε επιτέλους να βρούμε λύσεις. Κλείνοντας λοιπόν, να πω μια τελευταία κουβέντα. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου δεν θα πρέπει να αποτελέσει το τέλος, αλλά την απαρχή μιας διαδικασίας μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να δεσμευτούμε εμείς το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και το Εθνικά Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Δύσκολα θα σεβαστούμε το χρόνο από ό,τι φαίνεται, οπότε πρέπει να είμαι όλο και πιο περιοριστικός γίνεται ο κύριος Λακκουά από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Εξ ονόματος του Βελγικού Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας πω ότι και εμείς ψηφίσαμε μια απόφαση για τον καθορισμό του βελγικού στρατεύματος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καλό θα είναι να το κάνουν και οι άλλες χώρες. Εγώ βλέπω εδώ την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει η Γαλλική Γερουσία σαν παράδειγμα. Τώρα για τον προγραμματισμό. Κύριε Αρνούτ, επιμείνατε στον ανεφοδιασμό εμπτήση και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ έχουμε και το θέμα της ανανέωσης των καταδιοκτικών μας που θα κοστίσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται των καταδιοκτικών αναχαιτιστικών αεροσκαφών. Ε, είναι αν θέλετε το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος. Αν αγοράσουμε τα F-35 ε, και όχι αυτό που μας συστήνεται εσείς, δεν ξέρω πώς θα καλύψουμε τις δαπάνες που θα προέλθουν. Γι' αυτό στρέφομαι σε εσά για να πω ε, πού βρίσκεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, Πολεμικού αεροσκάφους. Έγιναν προσπάθειες, έγιναν συζητήσεις, χάθηκαν τα πάντα προς το παρόν. Ε, μήπως πρέπει εν περιπτώσει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια για να σχεδιάσουμε ένα ευρωπαϊκό πολεμικό αεροσκάφος. Την τεχνική την ελέγχουμε και πετύχαμε με το Airbus γιατί όχι και εκεί. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Θα ήθελα όμως, σαν κοινοβουλευτικός αριστερός, να επιμείνω σε μια έννοια πολύ σημαντική που δεν περιλαμβάνεται στις παρουσιάσεις σας. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στον τομέα της άμυνας. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια χαρακτηριστικά της στρατιωτικής μας δυνατότητας και ικανότητας. Εγώ σαν αριστερός επιμένω στη συνδρομή σαν παράδειγμα στα θύματα μιας πολεμικής σύγκρουσης. Δεν βλέπω να φαίνεται κάποιο πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα στόλο σαν παράδειγμα νοσοκομιακών σκαφών τα οποία θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται ε, επιτόπου για να βοηθούν ε, ε, εκεί που χρειάζεται Συρία, Λίβανος κτλ. Έτσι θα συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την Ευρώπη της άμυνας, γιατί δέχονται οι πολίτες φυσικά τις δαπάνες για τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους και των γεωστρατηγικών τους συμφερόντων, αλλά και για την ανακούφιση των υπολείπων συμπολιτών τους. Σας ευχαριστώ, σεβαστήκατε αυτό το οποίο ε, ε, παρουσιάσατε στο σωστό χρόνο. Για τα νοσοκομιακά σκάφη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται ε, με μικρά γράμματα βέβαια στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την δυνατότητα που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει τέτοιου είδους σκάφη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μποζίνοβιτς, τον Κροάτη, ε, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς πώς πάνε τα πράγματα εδώ, δεν έχει το άλλο να πει ότι δεν ξέρει πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτιμώ τις προσπάθειες ε, που οδήγησαν στις σημερινές συναντήσεις. Το θέμα που μας απασχολεί έχει στρατηγική σημασία όχι μόνο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας αλλά έρευνας αλλά και της Ένωσης γενικότερα. Έχει σημασία η συζήτηση αυτή να τεθεί στο σωστό ευρύ νομίζω πλαίσιο. Η Κροατία ε, συμμετέχει στον προβληματισμό αυτό μέσω των ε, ερωτημάτων που θέτουμε και εμείς στη χώρα μου. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ αρκετά χρόνια πλέον και σαν ευρωπαϊκή χώρα αναγνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά είναι θέματα τα οποία χαίνουν προς το παρόν. Υπάρχει και μια πρόκληση μπροστά μας. Από τη μία υπάρχει μια σχετική έλλειψη ικανοποίησης για τα τεχνολογικά μέσα που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, από την άλλη υπάρχουν λίγοι αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να υποστηρίξουν μεγαλύτερες πολεμικές προμήθειες, στρατιωτικές προμήθειες στην παρούσα φάση. Για διάφορους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά αναμένεται από αυτά να εφαρμόσουν κάποια ευρωπαϊκά επίπεδα στον τομέα το στρατιωτικό. Αυτό βέβαια απαιτεί λήψεις μέτρων ε, σε εθνικό επίπεδο. ψηλότερες δαπάνες βέβαια στον τομέα αυτό σημαίνει μείωση δαπανών σε άλλους τομείς. Όταν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί βέβαια το πρώτο θύμα είναι η άμυνα. Είναι σαφές ότι η αλληλοεπίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των χρηματοδοτικών είναι κάτι το δεδομένο και μπορεί να προκληθούν κάποιες παρανοήσεις οι οποίες θα αποδοθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη γνώση για τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε και στον τομέα της άμυνας και στον τομέα της αμυντικής πολεμικής βιομηχανίας. Με άλλα λόγια τι θέλω να πω όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς λόγους, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την άμυνα από τις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ως εκ τούτου λοιπόν θα τελειώσω λέγοντας ότι είμαι πεπισμένος ότι η συνεισφορά της άμυνας δεν είναι μια πιθανότητα αλλά μια ανάγκη αναπόφευκτη. Να προσθέσω κάτι συγκεκριμένο εδώ. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι λιγότερες δαπάνες στον τομέα της άμυνας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κρίσης της οικονομικής, αλλά και λόγω μη ύπαρξη συμβατικών απειλών των χωρών μας. Και αυτό ακριβώς είναι ο καρπός βασικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κύριος Κόβατς. Ουγγρικό Κοινοβούλιο, κύριε Σκόβατ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σα συγχαρώ για τη διοργάνωση τη συζήτηση αυτή από πλευράς της ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Επιτροπή ε, Άμυνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το γεγονό ότι προσκαλέσατε τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια και θεωρώ ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται πιο πολλά εθνικά κοινοβούλια εδώ στο γύρο αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκυρία πριν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου στα τέλη του έτου. Νομίζω ότι τα πιο πολλά άτομα που εκπροσωπούνται εδώ, που εκπροσωπούν ε, εδώ εθνικά κοινοβούλια και ευρωπαϊκά κοινοβούλια γνωρίζουν ότι πολλά πράγματα πολλά εκκρεμή ζητήματα υπάρχουν στα οποία έχουν αντίθετη θέση σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία. Να σας διασφαλίσω όμως ότι σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον ε, της ε, Ουγγαρίας και η Δημοκρατική Αντιπολίτευση και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας συμφωνούμε ότι το μέλλον της ε, Ουγγαρίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Για να είμαι σύντομος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων κινούμαστε. Καταρχάς, ότι το ΝΑΤΟ και ο ηγετικό ρόλος ε, των ε, ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αναφέρεται ως την κλίδα ασφαλείας για το μέλλον της Ευρώπης και την ασφάλεια της Ουγγαρίας. Αλλά η Ευρώπη, ακόμα και τα μέλη που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να συμβάλλουν ε, το ότι τους αντιστοιχεί στην ασφάλεια και την άμυνα της Υπήρου. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον παγκόσμιο και καθολικό ρόλο και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο έντονος παραποτέ. Είμαστε υπέρ δίκαιης και αποτελεσματικής ε, κατανομής των ευθυνών, ανάλογα και με τις ικανότητες των δύο οργανωτήτων και του δυναμικού των δύο οργανώσεων. Γιατί το ΝΑΤΟ έχει στρατιωτικά μέσα και μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε διαχείριση κρίσεων, ιδιαίτερα ενόπλων συγκρούσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιο πολύ δυναμικό και οικονομική ικανότητα πρόληψης ένοπλων συγκρούσεων και να συνδράμει στην ε, ε, φάση μετά την κρίση, μετά την επιλήξη της κρίσης. Ύστερα, η άμυνα είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα και εκτείνεται πέρα από τις ε, στρατιωτικές δαπάνες η ΚΕΠΑ και η κοινή άμυνα θα ωφεληθούν ενδεχομένως από άλλα μέσα, εμέσως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα μέσα τα οποία κατευθύνονται προς τους γείτονές μας. Στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, η εταιρική σχέση στη Μεσόγειο, η εταιρική σχέση προς Αντολάς γιατί η σταθερότητα και η ασφάλεια στις γειτονικέ χώρες είναι τμήμα της ασφάλειας και της δικής μας επίρου. Προσφάτως, η Αραβική Άνοιξη το κατέδειξε αυτό με μεγάλη σαφήνεια και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αντιμετωπίζουμε και την ε, εταιρική σχέση με τις χώρες της Ανατολής. Ε, η σημασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αναπόσπατα, αναπόσπαστα τμήματα της ε, πολιτικής ασφάλειάς μας. Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε από την αραβική Άνοιξη να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν και εδώ θα κλείσω να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο, να καλέσω και τα Εθνικά Κοινοβούλια να ασκήσουν πίεση στις δικές τους κυβερνήσεις για να προωθηθεί περαιτέρω η ενοποίηση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Μάλιστα, να δώσω το λόγο στους συναδέλφους Αναγκόμες γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. this context of the... Στο πλαίσιο αυτό της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας των προϋπολογισμών, το να μιλάει κανείς για άμυνα σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για τη βιομηχανική βάση η οποία θα στηρίξει τη συγκεκριμένη άμυνα. Ελπίζω επιτέλους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πάρει την απόφαση και να απορρίψει τα λεγόμενα offsets τα οποία επικρατούν στον τομέα των στρατιωτικών προμηθειών διότι είναι η βασική πηγή θα έλεγα διαφθοράς. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δράσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε ορθολογικό επίπεδο αλλά δεν έχω και πάρα πολύ εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο σε αυτό. Ελπίζω πάντως ότι κατελάχιστον τουλάχιστον ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, δεν θα μειώσει οικονομικά τις αποστολές τις οποίες ε, αυτή τη στιγμή διεξάγουμε και θα, συνεχίσει, ε, θα συνεχίσει να συνεισφέρει. Βλέπουμε πώς λειτουργήσε το θέμα στο Μαλί. Η θαλάσσια διάσταση της ΚΕΠΑ θα υπογραμμιστεί ελπίζω και θα της δοθεί ε, περιεχόμενο. Βλέπουμε την πειρατεία στον κόλπο της Γουινέας, βλέπουμε τα τρομοκρατικά δίκτυα, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μεσόγειο, όπου είναι σαφές ότι απαιτείται μια πραγματική ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και βλέπουμε επίσης την διεύρυνση ε, της σύραγγας του Παναμά το 2015, κάτι το οποίο ανοίγει νέε δυνατότητες αλλά δημιουργεί και περαιτέρω κινδύνους. Και στα σύνορά μας βέβαια, όπου όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν, είναι η Λιβύη. Το θέμα αφορά όχι μόνο την ασφάλεια της Λιβύης, αλλά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η UBAM, η υπάρχουσα αποστολή στη Λίβια, αν δεν μπορέσει να μετατραπεί σε πλήρη αποστολή με συγκεκριμένες υποδομές στρατιωτικές και αστυνομικές που δεν υπάρχουν σήμερα στη Λιβύη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς τις πολιτοφυλακές να λειτουργούν τη χώρα. Και απαιτείται να υπάρξουν αλλαγές και στον τομέα της ασφάλειας, δικαιοσύνης κτλ. και οι σύμβουλοι από τις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές για να δώσουν οδηγίες υποτίθεται για τη βελτίωση της ασφάλειας της χώρας λειτουργούν σαν πλασιέ για την πώληση των, πολιτικών, ε, των πολεμικών εξοπλισμών της ε, κάθε χώρας στην οποία εκπροσωπούν. Τελειώνοντας θα αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο ήδη θίξατε, την ανθρωπιστική διάσταση. Η ανθρωπιστική αυτή διάσταση βασίζεται στο Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο και στην παγκόσμια τάξη δικαίου. Αυτό απαιτεί ότι στον τομέα σαν παράδειγμα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει εμείς να διαφοροποιηθούμε από άλλους συμμάχους οι οποίοι δεν σέβονται το δίκαιο και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σαφώς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίσκο από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω περισσότερο κάποιες ερωτήσεις, οδεύοντας προς το Συμβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου. Δεν ε, είναι στην ημερήσια διάταξη, θα έλεγα τα θέματα αυτά, αλλά αναπόφευκτα θα τεθούν και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει τα ε, πληροφορικά συστήματα στον τομέα της ασφάλειας, συστήματα κεφαλαιόδη για να διασφαλιστούν οι ισορροπίες σε επίπεδο στρατηγικών και να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά κάποιο τρόπο οι ασθένειες της Ευρώπης έχουν ήδη έρθει στην επιφάνεια. Έχουμε προβλήματα στον τομέα της κατασκοπίας, έχουμε στο προβλήματα στον τομέα των ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων και διαβετώ τι θα γίνει επιτέλους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Έχει την δυνατότητα, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια κοινή στρατηγική η οποία θα επιτρέψει να βεθούν εγγυήσει για την προστασία της κυριαρχίας μας. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την δυνατότητα να δημιουργήσει με τη σειρά της ε, κάποια κέντρα που να διασφαλίζουν ε, την κυβερνοασφάλεια. γιατί οι πληροφορίες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό είναι φυσικά πηγές ανησυχίας και δείχνουν το ευάλωτο των συστημάτων μας συλλογής πληροφοριών. Τα όργανα μας, οι ζωές μας και τα συμφέροντά μας στον τομέα των επιστημονικό και των στρατιωτικό φυσικά απειλούνται. Και γι' αυτό θα πρέπει να προστατευτούν με σωστότερο τρόπο από απειλές και από ενέργειες κατασκοπίας όχι μόνο από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών. Γιατί έχουν και άλλες χώρες οι οποίες συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ηνωμένε Πολιτείες. Και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και δημιουργεί καταστάσεις ιδιαίτερως ανησυχητικές. Τέλος. Ευχαριστώ και για να κλείσουμε ο κύριος Λαντσμπέργης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλά σημαντικά ε, σημεία αναφέρθηκαν εδώ. Αν θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για μια συνεκτική ε, συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τελικά ίσως μια, ένα συνασπισμός των προθήμων για να εργαστούν σε μια ομάδα αλληλεγγύης, ίσως Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας κοινέ δυνάμεις για πρόληψη επιθέσεων. Καμιά φορά αυτό το σχήμα χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, μέσα στα πλαίσια ε, των Ηνωμένων Εθνών της ασφάλειας. Βεβαίως πολλές φορές ε, υπήρχε βέτο για κάθε προσπάθεια συνασπισμού των προθύμων Ε, και θεωρούσαν ορισμένοι ότι ήταν παράνομο διεθνώς. Έτσι η Ρωσία και η Κίνα απέκτησαν ε, φωνή σημαντική για διεθνή θέματα. Η πίεση αυξάνεται. Τίποτα χωρίς εμάς. Η Ρωσία ε, και η Κίνα δεν ξέρω αν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της ΚΕΠΑ τότε ο συνασπισμός ε, των προθήμων ίσως ε, να μπορούσε να γίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε περαιτέρω ε, στρατηγικές ή να μην αναγγείλουμε δράσεις αν δεν έχουν εγκριθεί από την Ρωσία να θεωρηθούν παράνομες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για αυτές τις παρεμβάσεις είδα ότι υπήρχαν πολύ λίγες ερωτήσεις για τους ομιλητές και σκέφτομαι τον κύριο Λακρουά για τις δυνατότητες. Θα δώσω τον λόγο ε, και στον κύριο Μισιρόλιο, ο οποίος μας ακούει υπομονετικά εδώ και αρχικό χρόνο, αρκετό χρόνο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ασφάλειας, μελετών για θέματα ασφάλειας, που ίσως μας δώσει μια άποψη πιο συνθετική ε, για αυτό το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για να κλείσω μετά θα δώσω τον λόγο στην Κλοντ France Αγνού και στον κύριο Ποπόφσκι που θα απαντήσουν ε, στις ε, ερωτήσεις ε, και θα συμπεράνουν. Δεν νομίζω ότι εγώ θα δώσω συμπληρωματικές πληροφορίες στο τέλος της συνεδρίασης να προσπαθήσω να κάνω μια σύνθεση της σημερινής συζήτησης και άλλων συζητήσεων στο παρελθόν τόσο εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο και σε ορισμένα εθνικά κοινοβούλια που με κάλεσαν για να κάνω σύντομες παρουσιάσεις. Θα περάσω στα αγγλικά τώρα. Λέχθηκε σωστά ότι η επιλογή του Προέδρου Φαντρομπόη να περιλάβει συζήτηση για άμυνα το Δεκέμβριο ήταν ένας κίνδυνος που ανέλαβε και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο και υπό το φως της συζήτησης που είχαμε μέχρι τώρα και σήμερα και προηγουμένως ε, νομίζω ότι αυτό το στίχημα πλήρωσε. Αν δείτε το θέμα της ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη πριν μερικούς μήνες και δείτε τι συνέβη, τι παρήχθη, τι δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών και μέχρι τώρα υπάρχει ήδη μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει ένας υψηλός βαθμός σύγκλησης και κονσένσους γενικής συνένεσης για ορισμένα επίγοντα θέματα που επισημάνθηκαν τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα Εθνικά Κοινοβούλια και από την κοινότητα των εμπειρογνωμόνων του οποίου είναι μέλος του Ινστιτούτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κονσένσους και σύγκληση σχετικά με την αξιολόγηση της γενικής κατάστασης, η ψαλίδα ανάμεσα στην άνοδο των ε, απειλών των προκλήσεων ε, για την Ευρώπη και από την άλλη μέρα την μείωση των δημοσιονομικών πόρων και την μείωση των πολιτικών πόρων σε σχέση με την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, προθυμία συντονισμού και αν εξετάσετε προσεκτικά τι έχει παραχθεί τόσο από τα όργανα όσο και από ανεξάρτητα think tank και ερευνητικά κέντρα, θα έλεγα ότι υπάρχει μια αξιολόγηση ρεαλιστική του τι μπορεί να επιτευχθεί το Δεκέμβριο και ίσως και μετά υπάρχει μια, μια ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης των πραγμάτων, διαθεσίμων, πόρων, κονσένσους που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Και αυτό είναι ήδη ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα ενεργητικό βεβαίως δεν αναπόκειται σε μένα να αξιολογήσω ποια θα είναι τα τελικά συμπεράσματα του Δεκεμβρίου, αλλά η διαδικασία μέχρι τώρα συνέβαλε σε ένα δυνητικά θετικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι μέρος του αποτελέσματος αποτελέσματος. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα αρκετά δύνατο το οποίο θα πρέπει να διαβιβάσουμε στους ηγέτες. Υπάρχει ένα σημείο υπό το φως της συζήτησης που θα ήθελα να επισημάνω. Το consensus, η σύγκληση. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες διαφοροποίησεις για το πόσο γρήγορα και πόσο μακριά θα έπρεπε να πάει ο συντονισμός και η ολοκλήρωση, αλλά υπάρχει μια σύγκληση σχετικά με τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν μέχρι ενός ορισμένου βαθμού. Αλλά σύνδεσμος που λείπει εδώ είναι η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη συζήτηση. Δεν συμφωνώ ότι οι, συζή... οι πολίτες έχουν ε, συμμετάσχει με πάθος σε αυτή τη συζήτηση. Ίσως, ε, ίσως δεν υπάρχουν τα μίντια. Αλλά αν δείτε τις ε, σφιγμομετρήσεις όχι μόνο των τελευταίων μηνών αλλά και ετών και το Ινστιτούτο δημοσίευσε μια έκθεση μας εκπλήσει το γεγονός ότι από τη μία πλευρά στον κατάλογο των πηγών ανασφάλειας για τους πολίτες συγκριτικά οι πηγές ανασφάλειας που μπορούν να αντιμετωπιστούν με στρατιωτικά μέσα έρχονται τελευταίες. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ενδιαφέροντος για το πώς οι στρατιωτικοί πόροι θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια. Αλλά η ανασφάλεια γενικά αυξάνεται στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι ότι συνεχώς συνεπώς ε, με την πάροδο των ετών οι πολίτες απαντάνε ναι όταν θέλουν περισσότερη κοινή δράση στην διεθνή σκηνή, περισσότερο ακτιβισμό από μέρους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσεις ανθρωπιστικές, πολιτικές και ασφαλείας γύρω από την Ευρώπη και παγκοσμίω, αλλά παντούνε συνεχώς όχι όταν τους ζητούμε αν θέλουν να αυξηθούν οι πόροι για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Αυτός είναι ένας κρίκος που λείπει και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν είναι αληθές ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Όταν έχουμε κρίσεις και η Συρία πριν από μερικούς μήνες είναι ένα παράδειγμα, αντιδρούν και πολύ συναισθηματικά αλλά ως προς τις απαντήσεις που θέλουν να έχουν από τους πολιτικούς δεν είναι αυτές που θέλουν οι πολιτικοί. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι τελικά ένας αριθμός κοινοβουλίων αποφάσισαν κατά της στρατιωτικής επέμβασης, ίσως αντικατοπτρίζει την άποψη των πολιτών. Υπάρχει μια κόποση μεταξύ των Ευρωπαίων ως προς τις εμπειρίες των τελευταίων ε, δεκαετιών που έδειξαν ότι η στρατιωτική επέμβαση αυτή καθεαυτή δεν συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Και ίσως Εκεί πρέπει να γίνει πρόσθετη εργασία από τους νομοθέτες, από τα think tanks, τις δεξαμενές σκέψεις, τους πολιτικούς ηγέτες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προβληθεί περισσότερο αυτό το θέμα για να πιστούν οι πολίτες για την χρησιμότητα των όσων συζητούμε σήμερα και στο παρελθόν για να αυξήσουμε τη δική τους ασφάλεια. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές περιπτώσεις που πρέπει να τους παρουσιάσουμε οικονομικά, ε, και πολιτικά και παγκόσμια θέματα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, ούτω ώστε να τον κάνουμε καλύτερο σε μια κατάσταση όπου υπάρχει αβεβαιότητα, αστάθεια και απροβλεψιμότητα. Ίσως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό όλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή σε αυτά σε σχέση με άλλες οργανώσεις και άλλες, άλλα όργανα. Μια διαδικασία όπου θα υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και των αποφάσεων πολιτικής και όπου θα υπάρχει και υλοποίηση των συμπεφωνημένων αποφάσεων. Ίσως το τελευταίο μέρος της πρωτοβουλίας που απαιτείται τις τελευταίες εβδομάδες πριν από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να δείξουμε σαφώς απέναντι στους πολίτες πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια και η άμυνα, ότι υπάρχει μια διαδικασία ορθολογική με συνέχεια, ότι θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό που θα συμφωνηθεί. Υπάρχουν ε, διαβουλεύσεις που παρουσίασαν ε, διάφοροι οργανισμοί εδώ, υπάρχει μια ευρύτατη συζήτηση που ενισχύει το θέμα και θα πρέπει όλα αυτά να ενισχυθούν ούτως ώστε η ευρωπαϊκή άμυνα ε, να γίνει ε, πιο σημαντική και επικοδομητική για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήσουν πάρα πολύ συνοπτικός και συνθετικός. Κλοντ Φρανς για να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες που τέθηκαν και για ένα γενικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ, Αρνό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αναφέρθηκαν σημαντικοί τομείς από πάρα πολλούς από εσά και που πρέπει να συζητηθούν στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων εξάλλου αναφέρονται στην έκθεση της κάθε Άστον η θαλάσσια ασφάλεια όπως είπε η κυρία ε, Γκόμες και Κοπά το θέμα εξάλλου των πλοίων νοσοκομείων μπορεί να αποτελέσει ένα θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί μέσα στα πλαίσια της θαλάσσιας ασφάλειας. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έχουμε ένα δίκτυο ανάμεσα στους στόλους που μπορούν να ε, αλληλεπιδράσουν στα πλαίσια Μαρσούρ και για να εξασφαλίσουν μια ασφάλεια θαλάσσια μέσα στα πλαίσια των όσων κάνει γενικά η Κομισιόν για την θαλάσσια ασφάλεια. Ο κύριος Γκαλέρ ανέφερε τα θέματα τυποποιήσεως και επιστοποίησης και νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα ουσιαστικό το οποίο παρά το τεχνικό χαρακτήρα του ε, μπορεί να αναδειχθεί σημαντικό με τα παραδείγματα και να συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε εντολή μας ανατεθεί. Το θέμα της ενέργειας. Μιλήσατε πολύ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός προτείνει στοιχεία έχοντας πλήρη συνείδηση ότι είναι μια συμβολή σε μια προσπάθεια πιο συνολική στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία στον κυβερνοχώρο. Απαντώντας τον κύριο Κλίσσας, ε, είναι ουσιαστική αυτή η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και υπάρχει τώρα ε, με το ACT ε, υπάρχει μια συνεργασία συνεχής για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν για το sharing, ε, pooling and sharing και το smart defense. Ανέφερε κάποιος άλλος Έχουμε το ΝΑΤΟ που είναι ε, ίσως ε, καθαρά στρατιωτικός οργανισμός ενώ εμείς ασχολούμεθα ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεροχή των αρχών του δικαίου Βεβαίως όταν ασχολούμεθα με τον ανεφοδιασμό με εν πτήση και τα remote ε, piloting systems, τα drones, ε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, τα εξαποστάσεως πλοηγούμενα συστήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι για δυνατότητες ε, καθαρά στρατιωτικές υπάρχει συμφέρον να έχουμε συνέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένω πάνω στο γεγονός ότι πρόκειται για δυνατότητες ε, που ε, αναπτύσσουμε χρησιμοποιώντας τα μέσα ε, της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, αλλά είναι τα μέσα που έχουν τα κράτη και που θέτουν στη διάθεση του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα του κυρίου Λακρουά για τα αεροσκάφη. Έχουμε τρία αεροσκάφη συν τα αμερικανικά. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε τρία μαχητικά ρεσκοφκάφη. Το Rafale, Eurofighter και έχουμε επιπλέον το F16, το F35. Ε, βεβαίως, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχουμε μια μελέτη για τα εναέρια συστήματα του μέλλοντος που αναφέρονται στο θέμα αυτό και θα περάσουμε στη δράση ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί πολιτικά από τα κράτη-μέλη. Η ελπίδα μου, αν μπορώ να πω κάτι προσωπικό, είναι ότι υπάρχει ίδια προσέγγιση όπως και για τα drones, τα μια επανδρομένα. Ε, υπάρχουν ε, εξοπλισμοί τους οποίους αγοράζουμε και βάζουμε από κοινού τα μέσα ρεαλιστικά και εργαζόμαστε στο το δυνατόν περισσότερο στην αρχή της φάσης για το μέλλον και για να έχουμε προγράμματα ευρωπαϊκά στο μέλλον. Σχετικά τα θέματα για το Eurogroup, για ένα Eurogroup και την, ε, μια μόνιμη δομημένη συνεργασία, αν, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, πολλοί με άκουσαν να κάνω αυτή τη παρατήρηση, είναι ότι η καλή έκπληξη της ΚΕΠΑ είναι ο ρόλος ε, των μικρών και μεσαίων κρατών μελών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ε, Ποιος γίνεται επικεφαλής για πολλά από τα προγραμματά μας είναι Φινλανδία, είναι η Εστονία, η Ιρλανδία για την εκπαίδευση, την Ναυτική, Αυστρία για πάρα πολλές από τις δραστηριότητές μας νομίζω οι κάτω χώρες, μιλάω και για μεσαίες χώρες, για την ανεφοδιασμό εμπτήση, ε, Νομίζω ότι όλα θα είναι εφικτά σε ομάδες περιορισμένες όταν θα υπάρχει εκπαίδευση των, στις μεγάλες χώρες και εδώ έχουμε πολύ περιθώριο ανάπτυξης ώστε τα μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξουν αυτό το ρόλο, να μπορούν να παρεσύρουν του άλλους. Ε, να κάνουν τους άλλους να είναι σε θέση να δράσουν. Αυτό περιμένουμε από τις μεγάλες χώρες, να παρασύρουν τις άλλες, διότι η νομιμότητά τους θα εξασφαλιστεί από τον ρόλο που θα παίξουν ε, δίνοντας ε, στους άλλους ε, την δυνατότητα να δράσουν με δυνατότητες πιο απαιτητικέ και με γνώσεις επιστημονικές και ανεφοδιασμό εμπτήση. Αυτό κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε με το πέρασμα του χρόνου αλλά και εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουμε ένα μέρος του φορτίου και θα κλείσω λέγοντας ότι το ίδιο το περιμένουμε και στον βιομηχανικό τομέα. Άκουσα τις ε, παρατηρήσεις ότι έχουμε δύο Ευρώπες, αυτοί που έχουν μεγάλες βιομηχανίες εθνικές και αυτοί που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ λίγες βιομηχανίες. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάποιος που δεν έχει καθόλου βιομηχανία και πολλές είναι διτές, διπλής χρήσης και ε, δεν, τα αντισταθμιστικά μέτρα βεβαίως είναι παράνομα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει μια θέση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νεοφερμένους στις βιομηχανικές δυνατότητες, στην αλυσίδα εφοδιασμού, στα αποκοινού προγράμματα και για να υπάρχει μια μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτούς που δεν είναι τόσο παλιοί, δεν είναι με τον ίδιο τρόπο και για τις μικρομεσές και αυτό είναι που μπορούμε να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βρουν έναν τρόπο ούτως ώστε ο καθένας να έχει ενδιαφέρον και συμφέρον για την παραγωγή και την απασχόληση στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ την Κλοντ Φρανς, ο κύριος Ποπόφσκι για να κλείσει. Η συζήτηση αυτή έδειξε για μια ακόμη φορά ότι οι συζητήσεις που γίνονται για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα θα πρέπει να ειδωθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στα πλαίσια δηλαδή της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι το σαφές και είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται στον τομέα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Έτσι θα μπορέσουν να εμπλακούν ακόμα περισσότερο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη συζήτηση αυτή. The of the High Βλέπετε στην έκθεση της ε, υπάτου εκπροσώπου ότι δεν προτείνει την δημιουργία νέων δομών και δεν διεκδικεί νέες αρμοδιότητες. Αυτό είναι συγκεκριμένη επιλογή. Εμείς δεν θέλουμε να αρπάξουμε οι εσδήποτε αρμοδιότητες. Απλά θέλουμε να προωθήσουμε την σύγκληση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Απαιτείται, ε, θα έλεγα, περαιτέρω δράση στον τομέα της συνεργασίας των Ευρωπαίων και σε σχέση με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και σε σχέση με τους προγραμματισμούς τους εθνικούς υπήρξαν συγκεκριμένες παραπομπές στα θέματα αυτά στην έκθεση της κυρίας Άστον. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σώμα το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό στον τομέα της άμυνας. Όχι, αλλά θέλουμε να υπάρξει διασύνδεση στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα με τις αποφάσεις για την ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων που λαμβάνονται κατά καιρού σε εθνικό επίπεδο. Θα συμφωνήσω επίσης με αυτό που είπατε ότι η ΚΕΠΑ είναι τμήμα γενικότερα της εξωτερικής πολιτικής, έτσι δεν είναι, και των εξωτερικών σχέσεων κατά συνέπεια. Είναι ένα από τα βασικά μέσα λοιπόν τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σαν ένωση, μαζί με άλλα, όπως η αναπτυξιακή πολιτική και οι διπλωματικές σχέσεις. Παραμένει το θέμα της πρόκλησης της έλλειψης της κοινή αντίληψης για ορισμένα πράγματα. Αναφερθήκατε ήδη σε αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές εκκλήσεις για μια νέα στρατηγική. Προσπάθησα να δώσω απαντήσεις στον τομέα αυτό λέγοντας ότι εμείς θέλουμε τη διαδικασία του αντικατοπτρισμού αυτού του οποίου γίνεται στην Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο. δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνουμε την κατάληξη αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες νέες μορφές απειλής οι οποίες εμφανίζονται οξύτατες μερικές φορές και που προκαλούν το κοινό, το ευρωπαϊκό. Η θαλάσσια ασφάλεια σαν παράδειγμα, βλέπουμε τι γίνεται στη Λαμπεντούσα, βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Αν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις νέες ε, απειλές, τότε θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας στο ευρύτερο κοινό. Για μικρή αναφορά τώρα στη χρήση των ικανοτήτων και πάγια ανθρωπιστικούς λόγους. Θα το αντιστρέψω λέγοντας ότι μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μορφές στρατιωτικών ικανοτήτων για ανθρωπιστικούς λόγους γενικά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η θαλάσσια αποστολή Αταλάντα η οποία ξεκίνησε παρέχοντας ασφάλεια στο πρόγραμμα παράδοσης τροφίμων στην Σομαλία και είναι αναπόσπαστο τμήμα της εντολής την οποία αυτή τη στιγμή διεξάγουμε. η χρηματοδότηση των αποστολών και πας το οποίο ε, αναφέρθηκε η κυρία Γκόμες. Έχει ήδη γίνει εν μέρη συζήτηση αυτή. Δεν υπάρχει συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την δημιουργία πιθανώς ε, μιας νέας δομής. Απ' την άλλη θα προχωρήσουμε σε μια επανεξέταση του μηχανισμού του ισχύοντος το 2015 και αυτό θα είναι μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών αποστολών αλλά να μην αγνοούμε την μη στρατιωτική διάσταση η οποία σήμερα δεν ήταν πάρα πολύ παρούσα. Και υπάρχει μια αναφορά στην έκθεση της ΥΠΑΤΟΥ λέγοντας ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε ίσως τους κανόνες οι οποίοι ορίζουν την χρηματοδότηση και την ΚΕΠΑ για πολίτες τετάρτης πλέον γενεάς. Αυτά είναι θέματα τα οποία ίσως γνωρίζετε. Ξέρετε τι, τι καταστάσεις συναντήσαμε στην α, Λιβύη και στο κέρας της Αφρικής με την αποστολή UCAPNEST. Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είχαμε μια, έχουμε μια στρατηγική, καθορίστηκε στις αρχές του 2013, έγινε μια ανακοίνωση πρώτα από την κυρία μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλήξαμε τον Ιούνιο. Η δομή αυτή ξεκίνησε παράλληλα με την νομοθετική πρόταση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός δικτύου οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων επικοινωνίας. Τώρα, για σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κοπά για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έγινε ήδη η συζήτηση αυτή με τα κράτη-μέλη. Είναι μια συζήτηση η οποία θα επιτρέψει την χρήση σαν παράδειγμα των μη χρησιμοποιημένων μέχρι τώρα δυνατοτήτων. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και ε, παραμένουμε, αναμένουμε αν θέλετε σε κάποιες περαιτέρω εξελίξεις τώρα για την επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς όμως γιατί τα θέματα αυτά συνδέονται με το θέμα της εθνικής κυριαρχίας θα ήθελα να πω ότι η επικοινωνία είναι κάτι το βασικό για όλους, όχι μόνο για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για το κοινοβούλιο αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η ασφάλεια και η άμυνα είναι σημαντικότατα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις ε, ήταν πυκνές, ήταν σαφείς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε ως εδώ για τη συνάντηση. Θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ προσοχή τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν στο Συμβούλιο και το ίδιο το Συμβούλιο. Θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούμε στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής διάσκεψης που θα γίνει υπό ελληνικής προεδρίας τον επόμενο Απρίλιο. Με αυτή την αφορμή θα έχουμε την δυνατότητα να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, ελπίζουμε να υπάρξουν αποτελέσματα, αν και όλοι συνειδητοποιούμε βέβαια ότι πρόκειται για την αρχή πλέον μιας διαδικασίας η συνοδεία αν θέλετε των μέτρων που θα εφαρμοστούν μεσοπρόθεσμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει. Όπως έλεγε ένας από τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των κρατών μελών δεν θα πρέπει η συνάντηση αυτή να είναι απλά μια άλλη συνάντηση πριν την επόμενη σε πέντε χρόνια. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε με συντονισμένο τρόπο και δεν θα πρέπει να μας ξεπεράσουν ε, τα πράγματα και η κρίση η οποία αυτή τη στιγμή μας απειλεί. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τις ομιλίες σας, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που τακτικά μας επισκέπτονται και ευχαριστώ και για τα, μέλη που ήρθατε εδώ σήμερα. Κλείνω λοιπόν τη συζήτηση λέγοντας ότι υπάρχει ένα, ένα μπουφέ βγαίνοντας από την ε, αίθουσα.